Καλησπέρα σε όλους. Μπορούμε να αρχίσουμε. Έχουμε το σχέδιο ημερήσια διάταξη, το οποίο το πήρατε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 8 πρώτου του 2010 και θα ήθελα να σας θυμίσω πιο συγκεκριμένα ότι όσον αφορά το 9, δηλαδή ε, ε, απαλλαγή 2008, Γενικός Προπολογισμός ΕΚ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όσον αφορά ε, τι ερωτήσει για την Όλαφ, θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Άρα θα συμμετάσχουν μόνο όσοι αναφέρονται στον κατάλογο που εδόθη στους συντονιστές από τη Γραμματεία και που εγκρίναμε πριν από λίγο στη συνεδρίαση του Προέδρου με τους συντονιστές. Οι γλώσσες αναφέρονται στο 2, 3, 1 ε, μεταδίδεται απευθεία από το διαδίκτυο η συνεδρίαση και πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να ευχαριστήσω την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου της Καταλωνίας και πιο συγκεκριμένα της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού του Κοινοβουλίου της Καταλωνίας. Τους ε, ήθελα λοιπόν να τους χαιρετήσω όλους, ε, εγκάρδια. Όπως αναφέρεται στις ε, πληροφορίες που έδωσε από τη Γραμματεία, ο κύριος Σόλ, ε, διευθυντής ε, του προπολογισμού ε, του ε, Κοινοβουλίου και η κυρία Φραντσέσκα Γκουαρτιόλα, που είναι πάλι επικεφαλής αρμόδιας υπηρεσίας στο Κοινοβούλιο της Καταλωνίας και εξ ονόματο τη Επιτροπή ε, Ελέγχου Προπολογισμού, ο κύριο Κόλλο, πρώην αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον οποίο θέλω να χαιρετήσω ε, ολόθερμα εξ ονόματο τη Επιτροπή μα. Κύριο Στιάνο επίση, ε, ο οποίο είναι επικεφαλή του αρμοδίου τμήματο τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Θέλουμε επίση να χαιρετήσουμε την κυρία Ούρσουλα Μοϊκόφσκα, στην οποία τη ευχόμαστε κάθε επιτυχία στι εργασίε τη. Και θα ήθελα να μας υπενθυμίσει ε, η Γραμματεία ότι να πάρουμε τα έγγραφα μαζί γιατί θα γίνει η αλλαγή αίθουσα. Όσον αφορά τα πρακτικά συνεδρία συνεδρίασης 2-3 Δεκεμβρίου, τα πήρατε και αν δεν έχετε να κάνετε κάποια παρατήρηση, νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίθηκαν τα πρακτικά. Σας παρακαλώ. Ähm, e- Το μέρια, κύριε Πρόεδρε. Στο Υπάρχει ένα, ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε στους συντονιστές στο πρόγραμμα και τα πρακτικά λέγουν στο αγγλικό κείμενο ότι αυτή η κυρία Γκρέσλε δηλαδή είναι η συγγήτρια <clears throat> πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό άρα προφανώς πρόκειται για μία παράληψη και πρέπει να είμαστε πιο σαφείς Ωραία. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, θα ε, φροντίσουμε να διορθωθεί το σημείο αυτό. Και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πάμε στο πρώτο σημείο τη ημερήσια διάταξη, που είναι η απαλλαγή 2008, Γενικό Προπολογισμό ε, ε, ΕΚ, τμήμα 3, Επιτροπή. Σα θυμίζω ότι όσον αφορά την ακρόαση για το σημείο αυτό, έχουμε μία ώρα. Λάβετε το υπόψη σας λοιπόν και απευθύνομαι κυρίως ε, στα μέλη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ε, κατά διατύπωση των ερωτήσεών τους. Λοιπόν, όσον αφορά το σημείο αυτό, να δώσω πρώτα το λόγο στον, στον κύριο Άραλ Νόακ, εξ του Ελεκτικού Συνεδρίου. Είναι εδώ στην αίθουσα. Σας παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κύρια, κύριοι μέλη της Επιτροπής, κύριε ε, Αντιπρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε. Εγώ ε, θέλω να παρουσιάσω εδώ μία σύντομη ε, παρουσίαση ε, και σας ευχαριστώ για το χρόνο το οποίο μου δώσατε εν ονόματι του ελεγκτικού συνεδρίου για να αναφερθώ στο θέμα αυτό και στην ανταλλαγή απόψεων με τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη και με τον Επίτροπο Τοπότσνικ. Στο κεφάλαιο 7 του, ε, της ετησίας για το 2008 ε, το συνέδριο αναφέρεται στον έλεγχο του τομέα της ερεύνης που αντιπροσωπεύει περίπου 6% των συλλογικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ενώσης για το 2008. Το κεφάλαιο 7 αναφέρεται στην έρευνα και όντως ε, ε, περίπου 80% από τις δαπάνες οφείλονται στα προγράμματα πλαίσιο της έρευνας. Άρα το, η πλειοψηφία των πληρωμών που εξέτασε το ελεγκτικό συνέδριο αναφέρονται στα προγράμματα πλαίσιο και ιδιαίτερως προσωρινές και τελικές πληρωμές για τα προγράμματα 6 και ε, προκαταβολές για το πρόγραμμα 7. Ε, άλλα βασικά θέματα είναι ε, για το TEN-T και TEN-E και αντιπροσωπεύουν περίπου 12%. Ουσιαστικά λοιπόν πρόκειται για μία ε, κεντρική διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή η Επιτροπή πληρώνει τους ε, αποδέκτες χωρίς να παρεμβαίνουν τα, οι αρχές των κρατών μελών. Ο μεγάλος κίνδυνος για την νομιμότητα και την τακτικότητα των δαπανών στην έρευνα είναι ότι οι αποδέκτες φουσκώνουν τα έξοδα τα οποία είναι επιλέξιμα εις ε, τις δηλώσεις τους που υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για αποπληρωμή από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αν αυτό δεν προληφθεί ή διατυπωθεί ε, ή διορθωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια. Ε, σύμφωνα με την προσέγγιση του ελεγκτικού συνεδρίου η μελέτη βασίστηκε σε δύο βασικά θέματα καταρχήν δείγματα 150 πληρωμών και ε, μία αξιολόγηση των βασικών ε, σημείων του συστήματος ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνολικά τα αποτελέσματα του ελέγχου 2008 κατά πολλήν επιβεβαίωσαν τις ε, διαπιστώσεις του 2007 και του 2006. Το ελεγκτικό συνέδριο κατέληξε ότι οι πληρωμές για την έρευνα, για τη μεταφορά και την ενέργεια και για το, τη σχετική ομάδα πολιτικής για το 2008 ε, επηρεάστηκε από ένα ουσιαστικό ποσοστό λάθους μεταξύ 2 και 5%. Η ε, επιτήρηση και ο έλεγχος και τα σχετικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μερικώς ε, αποτελεσματικά για να εξασφαλίσουν την τακτικότητα των πληρωμών. Παρόλη αυτή την ε, κατάληξη το Συμβούλιο το συνέδριο αποφάσισε επίσης να αναγνωρίσει τις προσπάθειες που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει τα συστήματα ελέγχου και να απλοποιήσει ε, τις διατυπώσεις χρηματοδοτήσεως και αυτά θα εφαρμοστούν ε, ε, τον χρόνο εργασίας της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής η βασική, τα βασικά είδη των ε, λαθών τα οποία μπορούν να αξιολογηθούν ε, φαίνεται να είναι η υπερβολική δήλωση των επιλεξίμων στοιχείων κόστους ιδίως ε, κόστη προσωπικού και έμεσα κόστη. Όπως και το 2007 υπήρχαν δηλώσεις μειώσεις κόστους που πάντοτε ε, που συχνά συνοδεύονταν από ένα πιστοποιητικό ελέγχου και ε, για το πρόγραμμα 7 σχεδόν όλες οι πληρωμές ήταν προκαταβολές και δεν διαπιστώθηκαν λάθη. Στην μελέτη της αποτελεσματικότητας των συστημάτων το συνέδριο βασίστηκε στο πρόγραμμα πλαίσιο 6 στο οποίο οι πληρωμές ε, είχαν οδηγήσει στα βασικά λάθη και ε, διαπιστώσαμε ότι η η έλεγχη των παραστατικών ήταν ικανοποιητική αλλά η ε, επιτόπιη έλεγχη δεν ήταν τόσο αξιόπιστη και ε, το συνέδριο διαπίστωσε λάθη σε 43% των πληρωμών τις οποίες εξέτασε. Πράγμα το οποίο μειώνει την ε, βεβαιότητα η οποία προσφέρεται από τα βασικά συσχεία του συστήματος ελέγχου. Το άλλο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βελτιώσει πάρα πολύ τη στρατηγική της ε, για τους ελέγχους εκ των υστέρων και ε, ιδίως ε, όσον αφορά την εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφοριών τα οποία βελτιώνουν τον συντονισμό μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων Ερεύνης. Εάν μπορώ δηλαδή να σας το εξηγήσω με απλά λόγια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξε θύμα της επιτυχίας της, διότι υπήρχαν πάρα πολλά μη επιλέξιμα στοιχεία κόστους που έπρεπε να καλυφθούν στην αρχή του 2008. Το σύστημα των κυρώσεων το οποίο ε, εφαρμόστηκε στην αρχή αρχή του προγράμματος πλαισίου 6 δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί και τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πολλές προόδους όσον αφορά το θέμα των καθυστερημένων πληρωμών. Ε, καταλήγω με τις συστάσεις. Δηλαδή, ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ελεγκτικό συνέδριο ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρήσει αυστηρούς ελέγχους, ιδίως για να βελτιώσει την αξιοπιστία των πιστοποιητικών ελέγχου και ε, επιζητώντας ε, μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή της ε, στρατηγικής ελέγχων εκ των υστέρων για να υπάρχουν έγκαιρες προσαρμογές και όπου αναγκαίο να εφαρμόζονται κυρώσεις. Ελπίζουμε ότι εις το μέλλον θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο συνολικές ε, πληρωμές ε, και μία καταποκοπή τιμή για τις ε, έμεσες δαπάνες. Θέλω τέλος να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας προσπαθώντας να επιτύχουμε ένα καλύτερο σύστημα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε τώρα τους δύο επίτροπους. Ε, και θα έλεγα πρώτα να δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο Ποτότσνικ εάν θέλει να τοποθετηθεί και σε σχέση με αυτά που ακούσαμε από τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου και συνέχεια να δώσουμε το λόγο ε, στον εισηγητή, τον κύριο Ριβεράσκη. Έχετε το λόγο, Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε αντιμαγκίστη, αγαπητή αντιπρόεδρη, αγαπητέ Δ. αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, συνάδελφοι. Σήμερα είμαι εδώ για να απαντήσω στις παρατηρήσεις στην έκθεση του Συνεδρίου του 2008 και σε ερωτήσεις των βουλευτών σχετικά με την έκθεση. Το πρώτο που θα ήθελα να σας τονίσω είναι το ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφωνία μεταξύ της Κομισιόν και του Συνεδρίου, μεταξύ εμού και του δόκτωρος Νόακ. Συμφωνούμε με την ανάλυση των δυσκολιών και οι έλεγχοι μας και των μεν και των δε δείχνουν πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το Ελληνικό Συνέδριο αναφέρει σημαντική βελτίωση στη διαχείριση, αλλά επίση επισημαίνουμε ότι η κατάσταση δεν είναι ακόμα απόλυτα ικανοποιητική. Το ίδιο λέει και η Κομισιόν. Πιθανότατα θα είναι η τελευταία ακροασίμω ε, επιτρόπου έρευνα και δεν ε, αφήσαμε στον πειρασμό να αναλογιστώ τι βελτιώσει που έγιναν στα τελευταία χρόνια στη διαχείριση του Ταμείου Έρευνα. Πολλοί από εσάς είστε νέοι ευρωβουλευτές, γι' αυτό θα ήθελα να, τα, να σας δώσω μερικά περισσότερα στοιχεία. Το 2006 ε, εντοπίστηκαν ποσοστά ασφάλματος 8% και ε, ότι η πολιτική ελέγχου δεν ήταν αποτελεσματική. Τα συστήματα υποπτίας και ελέγχου εφεωρήθησαν από το συνέδριο ανεπαρκή σε σχέση με τον κίνδυνο επιστροφής υπερβολικού στοιχείου κόστους. Η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού σωστά επισήμανε αυτές τις ανεπάρκειες, ατέλειες και προσπάθησε να βελτιώσει την κατάσταση. Από το 2006 και με τη δική μου βοήθεια εισαγάγαμε σημαντική βελτίωση στη διαχείριση με νέα στρατηγική ελέγχου με στόχο το υπολοιπόμενο ποσοστό λάθος να το φέρουμε κάτω από το 2% σε πολυετή βάση μέχρι το τέλος χρονικό πέρας της εφαρμογής κάθε προγράμματος πλαισίου. Αυτό απαιτούσε μεγάλη αύξηση των ελέγχων από 42 ελέγχους το 2006 σε 1084 ελέγχους το 2008. Σημαντικοί πόρια έπρεπε να μετατοπιστούν για να το πετύχουμε αυτό, αλλά το θεωρήσαμε αναγκαίο. Επίσης, φροντίσαμε ο στόχος των ελέγχων να είναι προς πιο μεγάλους και πιο επικίνδυνους δικαιούχους, έτσι ώστε να έχουμε πιο αποδοτική και μεγιστοποιημένη κάλυψη. Επίσης κάναμε και προβολή των ελέγχων. Δηλαδή όταν ένας δικαιούχος απεδείχθη ότι συστηματικά υπερέβαλε τις δαπάνες, ε, τότε ζητήσαμε ανάκτηση των ποσών για όλα τα συμβόλμα, ακόμα και αν δεν είχε γίνει έλεγχος. Βέβαια, καλό θα είναι να αποφεύγουμε τα λάθη εντελώ παρά να τα εντοπίζουμε και να τα διορθώνουμε μετά. Και ο πιο καλός τρόπος να αποφύγει κανείς το σφάλμα είναι να έχει απλούς κανόνες. Και δίνουμε συνεχώς αυτή τη μάχη να απλοποιήσουμε το σύστημα επιστροφής του κόστου, το FP7. Έχουμε ένα ταμείο εγγύησεων που μειώνει σημαντικά τους εκ των προτέρων ελέγχους. Μειώσαμε τα πιστοποιητικά ελέγχου σε δηλώσει κόστους. Έχουμε μια ενιαία, ενιαίο μέσο μητρώου ή καταγραφής. Και έτσι δεν έχουμε ανάγκη πολλών, πολλές φορές να έχουμε την ίδια πληροφορία. Και τέλος χρησιμοποίησαμε τους καταποκοπή συντελεστές και τα αποκοπή ποσά όπου ήταν αυτό δυνατόν. Με δύο εκτελεστικές υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν, απλουστεύσαμε τα πράγματα διοικητικά. Το πρεσμένο καλοκαίρι γίναμε αυτόνομοι. Και μόλις τότε είχαμε το πλήρες προσωπικό που χρειαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, πληρώνουμε πιο γρήγορα και τα συμβόλαια κλείνονται πιο γρήγορα. Για να έχουμε όμω ένα καλύτερο αποτέλεσμα στη στρατηγική του ελέγχου, ο στόχος θα πρέπει να είναι να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος και αυτό αναγνωρίστηκε από το ψήφισμα απαλλαγή του Κοινοβουλίου του 2007 και από την έκθεση του συνεδρίου. Αυτή η τάση συνεχίστηκε και το 2008 και το 2009 αν και ακόμα δεν έχουμε πετύχει τον τελικό μας στόχο 2%. Εξίσου σημαντική είναι η διαπίστωση ότι η στρατηγική ελέγχου μας είναι υγιής απευθυνόμαστε στου κινδύνους υπερβολικής δήλωση κόστου, του κινδύνου που ακριβώς επεσήμανε ο κύριος Νόακ. Είναι αναφυσβήτητο ότι τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σημαντική πρόοδος, αλλά θα πρέπει να κινηθούμε προς πλήρη εφαρμογή της στρατηγικής μέχρι το τέλος του 2010, που σημαίνει περισσότερη δουλειά, ιδιαίτερα σε δύο συγκεκριμένους χώρους. Αυτά επισημαίνονται και οι δύο στην ετήσια έκθεση του ε, συνεδρίου. Ανάκτηση, recovery και απλούστευση, simplification. Καταρχήν, ανάκτηση. Εδώ έχουμε δύο ιστορίες. Τις τακτικές ανακτήσεις και ε, ε, ανακτήσεις οι οποίες στηρίζονται σε χρονική προβολή, extrapolation. Σε σχέση με τις πάγιες ανακτήσεις συμβολέων που έχουν περάσει από έλεγχο, το ποσό ήταν σχετικά μικρό μέχρι το τέλος του 2008. Πάντως, το 2009 σημειώθηκε σημαντική πρόοδος και στο τέλος του χρόνου η Κομισιόν είχε διανακτήσει το 60% των οφειλόμενων ποσών σε σχέση με 30% που θα δείτε στην έκθεσή μας για το 2000, στην έκθεση του συνεδρίου για το 2008. Τώρα, όσον αφορά την διόρθωση συστηματικών λαθών με την χρονική προβολή Extrapolation το Κοινοβούλιο μας ζήτησε στην απαλλαγή του 2007 να μην επαναυπολογίζουμε τις οικονομικές δηλώσεις συμβολέων που είχαν κλείσει με βάση το FP6. Στις απαντήσεις που δώσαμε και σε μια επιστολή που έστειλα στον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής σας, ήμουν ασαφής. Όταν κάνουμε χρονική προβολή δεν ξαναυπολογίζουμε, διορθώνουμε εντοπισθέντα σφάλματα που είναι συστηματικά. Αν δεν διορθώσουμε αυτά τα σφάλματα, θα έχουμε πάγια σφάλματα περισσότερα εκ των υστέρων. Το Κοινοβούλιο επίση ζήτησε απλούστευση της διαδικασίας ανάκτηση με το ψήφισμα 17 Δεκεμβρίου 2009 στο σχέδιο Γενικού Προπολογισμού. Όπω σα είπε και ο κύριος Νόακ, είμαστε θύμα τη επιτυχία μα στην περίπτωση αυτή. Αυξήσαμε πάρα πολύ σημαντικά τα εντοπιζόμενα σφάλματα Φυσική συνέπεια αυτού είναι χρειάζονται πολλές διορθώσεις, που σημαίνει πολύ περισσότερες ανακτήσεις ποσών. Αυτό είναι μεγάλο διοικητικό βάρος και για την Κομισιόν και για τους δικαιούχους. Ιδιαίτερα αν προσθέσουμε και τις ανακτήσεις με βάση την χρονική προβολή προς το μέλλον. Πρέπει να πετύχουμε μια δύσκολη ισορροπία. Να αποφύγουμε διοικητικό βάρος, αλλά να έχουμε και το πιο μικρό δυνατό επίπεδο σφάλματος. Ε, λοιπόν, με ευχαρίστηση μπορώ να σας δηλώσω ότι η Κομισιόν πρόσφατα στις 15 Δεκεμβρίου ενέκρινε μια ανακοίνωση για την απλούστευση των ανακτήσεων που θα πρέπει να ικανοποιεί το αίτημα του Κοινοβουλίου. Και πιστεύω ότι πετυχαίνουμε τη σωστή ισορροπία. Η απλοποίηση αυτή δίνει τη δυνατότητα σε ένα καταποκοπή συντελεστή προκειμένου να οραστούν τα εκκρεμή χρέη και ορισμένα βάρη που με το προσωπικό όπως άμεση φόροι και οι κοινωνικές εισφορές πρέπει να θεωρούν ως ε, αποδεκτές, επιλέξιμες. Δεύτερον, η απλοποίηση. Τα μέτρα απλοποίησης ε, δεν έχουν λύσει βέβαια όλα τα προβλήματα μέχρι στιγμή. Στους προσεχείς μήνες θα υποβάλουμε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις, δυσκολίες. Πρώτον, μια ανακοίνωση προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την απλούστευση στη χρηματοδότηση της έρευνας. Την ετοιμάζουμε την πρόταση. Στηρίζεται σε πολύ μεγάλη διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους. Και θα ξεκινήσει μια μεγάλη διοργανική συζήτηση με νέες έννοιες για τη χρηματοδότηση της έρευνας όπως συστηματική εφαρμογή του καταποκοπή συντελεστή και καταποκοπή ποσών όπως πρότεινε το συνέδριο. Ε, ο Δ. Νόακ με ενθάρρυνε με αυτά που είπε. Οι έλεγχοι του συνεδρίου αναγνωρίζουν την ανάγκη καταποκοπή ποσών μέσων όρων και καταποκοπή συντελεστών που σημαίνει ότι να υπάρχουν σφάλματα σε σχέση με αυτούς τους συντελεστές, όχι με βάση το πραγματικό κόστος. Βέβαια, αν θέλουμε αυτή τα μέτρα πλήρους απλούστευσης να είναι αποτελεσματικά, θα πρέπει να συζητηθούν να συμφωνήσουμε στη μεθοδολογία εκ των προτέρων και ελπίζω η τεχνική ομάδα που έχουμε συστήσει μεταξύ των ελεκτών του συνεδρίου και των ελεκτών της Κομισιόν να συμφωνήσουν πώς θα κινηθούν στην πράξη. Και το δεύτερο μέτρο είναι πρόταση να εφαρμοστεί στην πράξη η έννοια του ανεκτού κινδύνου σφάλματος για δαπάνη έρευνας. Όσο πιο οι κανόνες, τόσο πιο λίγα τα λάθη. Τα τελευταία χρόνια Προσπαθήσαμε να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες και τους κανόνες. Αλλά στα πέντε χρόνια που ήμουν επίτροπος με, για, υπεύθυνος για προγράμματα έρευνας έμαθα ότι όλες αυτές οι βελτιώσεις είναι καλοπροαίρετες απαιτείται μια πιο ευρία προσέγγιση. Η έννοια του ανεκτού κινδύνου σφάλματος σε συνδυασμό με τα αποκοπή ποσά μέσους όρους κατά αποκοπή συντελεστές είναι μια σπουδαία ευκαιρία να απλουστεύσουμε την ερευνητική δαπάνη λαμβάνοντας υπόψη από τη μια την ανάγκη για υγιή διαχείριση της χρηματοδότησης της έρευνας και από την άλλη το κόστος ελέγχων. Στόχος μας θα πρέπει να είναι να έχουμε όρους που να είναι ελκυστικοί για τους ερευνητές να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να πάρουν μέρος στις κοινέ ευρωπαϊκές δραστηριότητες έρευνας. Υπεύθυνοι ερευνητέ που γνωρίζουν ότι η υγιής διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας και της ευθύνης είναι προς το συμφέρον τους. Και είδα ότι και το Ελεκτικό Συνέδριο και η Επιτροπή σα μα υποστήριξε σε αυτό τα τελευταία δύο χρόνια και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί. Βέβαια, η έννοια του ανεκτού κινδύνου σφάλματος δεν σημαίνει ότι γίνεται για να διευκολυνθεί μόνο η Κομισιόν. Ο διάδοχός μου που όπως ξέρετε είναι πρώην μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, έχει μεγάλη εμπειρία και είναι κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση αυτή, θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την ισορροπία αυτή όσον αφορά την έρευνα, την άνοιξη με το επίπεδο του ανεκτού κινδύνου λάθους, τις πολιτικές ανάγκες, τα ωφέλη της πολιτικής, τους εγγενείς κινδύνους και το κόστος ελέγχων και για την Κομισιόν και για τους διηγούς. είμαι σίγουρος ότι θα τον στηρίξετε, ότι θα την στηρίξετε, προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η απλούστευση και η χρηστή οικονομική διαχείριση. Ε, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ και μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου, η απλούστευση, η ευθύνη, η περιοδικότητα, η νομιμότητα, η καλή υπηρεσία για του ερευνητέ ήταν, είχαν προτεραιότητα στο έργο μου. Δέχομαι ότι δεν τα πέτυχα όλα όσα θα ήθελα, αλλά πιστεύω ότι από κοινού δημιουργούσαμε καλέ συνθήκε για σημαντικά βήματα και μέτρα που θα ληφθούν στο προσεχέ μέλλον. Η ανακοίνωση και η απλούστευση για την χρηματοδότηση τη έρευνα σύντομα θα την έχετε στα χέρια σα. Θα έχουμε την έννοια του ανεκτού κινδύνου στην έρευνα. Ετοιμάζεται και αυτό. Η τακτική αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και αυτό γίνεται. Όλα αυτά είναι σημαντικέ ευκαιρίε, Ιδεώδη ευκαιρίες που δεν θα πρέπει να τις χάσουμε. Επίσης, η επίγνωση του ότι πρέπει να εξυγχρονιστούμε στις μεθόδους μας. Θα έχω άλλο χαρτοφυλάκιο στο μέλλον, αλλά να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας, στην κοινή σας προσπάθεια για αυτό το στόχο. Τέλος, σας ευχαριστώ για το ανοιχτό σας πνεύμα, την επικοδομητική προσέγγιση, την επικοδομητική κριτική Φυσικά έχουμε διαφορετικούς ρόλους, σημαίνει και ιδέα. Πάντως συνεργαστήκαμε σε γνήσια εταιρική σχέση, εταιρική σχέση για καλύτερη έρευνα και για μια καλύτερη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Λιμπεράσκη που είναι ο εισηγητής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να σας πω ότι ήταν μεγάλη ευχαρίστηση για μένα ε, να ακούσω αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Νόακ και ο κύριος Ποτότσνικ. Εγώ πιστεύω ότι ε, κύριε Επίτροπε ε, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό, το οποίο ε, έγινε ε, σε σχέση με το πώς αναλάβατε στα καθήκοντά σας και το πόσο μάθατε μέσα από όλη αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Εδώ μιλάμε για ανεκτό κίνδυνο σφάλματος. Το σφάλμα σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Ο κίνδυνος είναι κάτι το οποίο το ε, διατρέχουμε κάθε μέρα. Αντί λοιπόν να μιλάμε για ανεκτό κίνδυνο σφάλματος, θα ήταν καλύτερο να μιλήσουμε για δικαιολογημένο ε, κίνδυνο σφάλματος. Δεν ακούγεται καλύτερα. Και αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και με βάση την εμπειρία σας. Και στη συνέχεια κύριε Πρόεδρε θα κάνω και μια δεύτερη ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι... Ναι, σε ευχαριστώ. Ε, αυτό το οποίο είπατε στον ορισμό σας είναι αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε και εμείς, προφανώς. Και συμφωνώ ιδιαίτερα ότι αυτή είναι η ουσία του ζητήματος το οποίο μας απασχολεί. Να σε εξηγήσω τώρα λίγα πράγματα, τα οποία ε, προσωπικά πιστεύω εγώ ε, πάντα όσον αφορά το ανεκτό, την ανεκτό κίνδυνο σφάλματος. Αν, αν, έχουμε το, το, το, το, σύστημα το οποίο έχουμε για όλα τα ε, προγράμματα πλαίσιο, 5, 6, 7, το οποίο στηρίζεται στα πραγματικά κόστη. Πρέπει να σα πω ότι το σύστημα αυτό είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Και αν έχουμε ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα, τότε καταλαβαίνετε ότι αν θέλουμε να, δούμε, να μειώσουμε τα, τα σφάλματα, το επίπεδο κόστους, αν θέλουμε να πέσουμε από το 8% στο 7%, είναι πολύ μικρότερο από ότι αν θέλουμε να πάμε το 3% στο 2%. Αυτό νομίζω είναι σαφές σε όλους. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο όπου θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να αντιμετωπίζουμε ε, με μια σοβαρότητα το ζήτημα και να πούμε εξακολουθούμε να μιλάμε για χρηστή διαχείριση. Και εδώ υπάρχουν δύο λόγοι για αυτόν τον ανεκτό κίνδυνο ή δικαιολογημένο κίνδυνο, αν θέλετε. Πρώτον, ε, το πραγματικό κόστος και το δεύτερο, η, η πολυπλοκότητα των κανόνων. Αυτό το οποίο ε, βρισκόταν στρατηγική για το πρόγραμμα πλαίσιο ε, το 6 και εκεί όπου δεν υπολογίσαμε καλά ε, αφορούσε τα μη συστηματικά επίπεδα σφαλμάτων. Είδαμε ότι το επίπεδο μη συστηματικών σφαλμάτων ήταν πολύ ψηλότερο από ό,τι είχαμε υπολογίσει στην αρχή. Κατά προσέγγιση, ωραία, 1,84 έτσι. Οπότε το κατά δεν έχει νόημα, δύο δεκαδικά χρησιμοποίησα. 1,84, άρα πολύ ψηλό. Λοιπόν, άρα αν θέλετε, ή μάλλον, αν εμείς, ε, ε, αν εμείς ή εσείς εξακολουθήσουμε να ακολουθούμε την, την οδό της πραγματικής απλούστευσης και απλοποίησης, για τα εφάπαξ ποσά, για, τις, ε, για τα καταποκοπή και αν κάνουμε σαφή διάκριση ανάμεσα στην απόκληση και στο σφάλμα, γιατί για μένα αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Απόκληση και σφάλμα. αν μιλάμε για τα εφάπαξ ποσά και τους μεσόρους. Αν αυτό γίνει σωστά, τότε είμαι σίγουρος ότι δεν χρειαζόμαστε αυτήν την έννοια του ανεκτού ε, κινδύνου σφάλματος. Αλλά με τα σημερινά πλαίσια, όπως έχουν τα πράγματα, νομίζω ότι όλα αυτά είναι αναπόφευκτα. Πιστεύω λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία ε, βρίσκονται στο στάδιο της ετοιμασία και ίσω το άμεσο μέλλον για μένα η καλύτερη προσέγγιση θα ήταν να συνδυάσουμε και τα δύο και να εμβαθύνουμε ε, στους μέσους όρους και τα εφάπαξ ποσά και από την άλλη να μιλάμε για τον δικαιολογημένο κίνδυνο σφάλματος όπως πολύ σωστά και εσείς είπατε ότι πρέπει να το ονομάζουμε. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ ε, κύριε Επίτροπε. Όσον αφορά αυτό το 43% των ε, υποθέσεων που ελέγχθηκαν και που ανέφερε και ο κύριος Νόακ, κατά την άποψή σας Επίτροπε, τι σημαίνει αυτό το ποσοστό. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση και θα μπορούσατε να εξηγήσετε, να μας εξηγήσετε το πώς κατά την άποψή σας το συνέδριο κατέληξε σε αυτό το ποσοστό σφάλματος. Και μέσα σε αυτή τη γενική ε, ατμόσφαιρα βελτίωσης δέχεστε αυτό το στοιχείο και αυτές τις εξηγήσεις ή μπορείτε να μας το εξηγήσετε παραπάνω. Μιλώ και αυτό το 43%. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, γιατί αυτά είναι τα γεγονότα. Το μόνο που θα μπορούσα να κάνω, να προσπαθήσω να σα εξηγήσω γιατί ε, συνέβη αυτό και γιατί δεν θα πρέπει να συμβεί στο μέλλον. Και να προσπαθήσουμε όλοι να μην συμβεί στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, έχουμε δύο λόγου που επίση είναι κρίσιμη σημασία. Το ένα έχει να κάνει με την περιπλοκότητα των κανόνων. Και το άλλο στοιχείο έχει να κάνει με το γεγονό ότι οι ελεκτέ είναι περισσότερο εξοικειωμένοι μερικέ φορέ με του εθνικού κανόνε και όχι τόσο με του Ευρωπαϊκού. Γιατί ο Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο των Πανεπιστημίων έκανε μια πρόσφατη μελέτη και έδειξε ότι υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά των χρηματοδοτικών κανόνων και των λογιστικών πρακτικών σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση η λύση για το πρόγραμμα πλαίσιο, για το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο, και εκεί βεβαίω είχαμε περισμένη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα, ήταν, το εξή. ήταν η εξή. Δώσαμε κατευθυντήριε γραμμέ για όλου του ελεκτέ, για τα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται από, το, από του εξωτερικού ελεκτέ. Και αυτά μπορείτε να δείτε σήμερα στο Κόρντι. Όσον αφορά το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, εκεί προτάθηκαν και ακολουθήθηκαν θεμελιωδέστερες αλλαγές. Πρώτον, πήγαμε στα λεγόμενα συμπεφωνημένα με βάση διαδικασίες. Οι ελεγκτέ δηλαδή συμφωνούν πάνω συγκεκριμένε διαδικασίε και αποφασίζει η Επιτροπή. Δεύτερον, πιστοποίηση μεθοδολογία υπολογισμού του κόστου ε, και τρίτον, το τρίτο πράγμα το οποίο κάναμε για να απλοποιήσουμε τα, ό, όλο αυτό το θέμα είναι ότι αυτά τα πιστοποιητικά ελέγχου ε, απαιτούνται μόνο για σχέδια άνω των 375.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ε, θέμα και αυτό το πρόβλημα που για να είμαι ειλικρινής είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο γεγονός. Γιατί εδώ μιλάμε ότι στην ουσία αμφισβητούμε το εκ των προτέρων, το προληπτικό τμήμα των ελέγχων, ενώ από την άλλη ε ε, ε, ε, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πίεση στους ελέγχους εκ των υστέρων. Ναι, Επίτροπε, αλλά στην ουσία, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής έρευνας, ε, πρέπει να δείτε εκεί τις ευθύνες σας. Δεν είσαστε ελεκτική υπηρεσία. Ο γενικός στόχος είναι η έρευνα. Αυτό είναι το χαρτοφυλάκιο. Κατά την άποψή σας, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πλησιάζουμε περισσότερο τις Ηνωμένε Πολιτείε στον τομέα της έρευνας. Δηλαδή η πολιτική που ακολουθούμε βοηθά τους ερευνητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ίσως έχει και νόημα να αντιμετωπίζουμε και να λαμβάνουμε έναν ανεκτό κίνδυνο εάν τελικά έχουμε κάποια ε, μεγαλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της έρευνας. Άρα με βάση την εμπειρία σας, το ξαναλέω, τι πιστεύετε ότι πετυχαίνουμε όλα αυτά τα χρήματα. To, to say... Το να ξέρουμε αν έχουμε προσεγγίσει τους Αμερικανούς ή όχι είναι κάτι δύσκολο. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε εισάγει ορισμένα από τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν και οι Ηνωμένε Πολιτείε και είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Όταν ε, αυτό εφαρμόστηκε ή στην Αμερική ε, αυξήθηκε η αποτελεσματικότητα της ε, Ευρώπης και οι Αμερικανοί μας κοιτούν πλέον σαν πιο σοβαρούς τους και αυτές, αυτούς τους απόϊχους έχω από την Αμερική. Ο ρόλος μας λοιπόν ουσιαστικά πρέπει να επικεντρωθεί στο να έχουμε την ε, καλύτερη έρευνα με τα καλύτερα αποτελέσματα για τα θέματα που μας καίνε. Ε, είτε μιλάμε για τον Ευρωπαίο πολίτη είτε για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αν με ρωτάτε λοιπόν ποια είναι τα σωστά βήματα για το μέλλον θα χρειαστεί ε, σαφώς απλοποίηση διότι ε, εάν μου δοθεί ευκαιρία ξέρω τι πρέπει να κάνω, θα το κάνω διότι δεν θα μας δοθεί άλλη ευκαιρία. Είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε και πιστεύω ότι τώρα είναι η η συγκυρία και γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι το γεγονός ότι έχουν αλλάξει τα στοιχεία ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν μιλάμε πλέον μόνο για τις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά και τους Ιαπωνέζους ούτως ή άλλως την Κίνα, τους Ινδούς και άλλους που αναπτύσσονται. Εάν λοιπόν ε, ε, τι τις δυνάμεις μας και υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα επιτύχουμε. Η προσπάθειά μου θα ήταν να αναστρέψω την φιλοσοφία των, της Γενικής Διευθύνσεως από τα προγράμματα εις ε, ένα ενιαίο ε, πρόγραμμα πλαίσιο με όλα τα ερευνητικά προγράμματα σαν σύνολο. Σας ευχαριστώ. Ε, κύριε Επίτροπε, ε, συμφωνώ ιδίως για την Κίνα και την Ινδία. Ίσως η Ινδία έχει περισσότερους φοιτητές πανεπιστημίου από ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο περίεργο και να μας φαίνεται. Αλλά μιλάμε για απλοποίηση. Ε, συστήματα καταποκοπήν πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να εφαρμοστούν χωρίς να αλλάξει το ισχύον σύστημα θα μπορέσουν δηλαδή να ενσωματωθούν στο σύστημα αυτό ή θα διαταράξουν πάρα πολύ ε, το ισχύον σύστημα. Δεν νομίζω θα το διαταράξουν διότι ουσιαστικά μιλάμε για χρηστή διαχείριση και οι ε, πληρωμές κατά αποκοπή δεν είναι άγνωστες στην Ευρώπη. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις είναι δύσκολο να εφαρμοστούν γιατί ξέρετε ότι οι διαφορές μεταξύ χωρών μπορεί να είναι ένα προς 10 και υπάρχουν ε, μεγάλα κενά. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ ακριβείς και πολλές ε, εργασίες θα πρέπει να βασιστούν σε μεθοδολογία όταν μιλάμε ε, για κατά αποκοπήν πληρωμές. Θα σας πω όμως ποιο είναι κατά τη γνώμη μου το βασικό πρόβλημα. Εάν, παραδείγματος χάρη, ε, ε, καταρτήσουμε ένα μέσο όρο και μετά μπορέσουμε να ελέγξουμε την απόκληση από το μέσο όρο και ελέγξουμε την απόκληση ε, διαμέσου των χρηστών και του τομέα θα πρέπει να υπάρχει μικρή απόκληση αλλά είναι μία απόκληση. Αν λοιπόν δούμε σε μεμονωμένες περιπτώσεις ότι η απόκληση ε, απέχει πολύ 30, 40, 50% κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται για λάθος αλλά απλώς διότι δεν, ότι δεν κοιτάξαμε μία μεμονωμένη περίπτωση σε, στη συνολική της ε, προοπτική και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα σωστός ορισμός να ξέρουμε ε, ποια είναι η απόκληση την οποία αν πρέπει να εξετάσουμε μεθοδολογικά και ποιο είναι το σφάλμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με πιο αυστηρά μέτρα, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή κατανόηση. Και ελπίζω ότι αυτό θα μπορέσει να επιτευχθεί στο νέο δημοσιονομικό κανονισμό και από πλευράς της Επιτροπής θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε ευρέως και με τα μέλη αυτής της Επιτροπής την ιδέα αυτή αλλά χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο του σκέπτεστε που έχουμε. Ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Βρισκόμαστε σχεδόν ε, ήδη στο φιλοσοφικό επίπεδο και φαντάζομαι ότι η φιλοσοφία πρέπει να είναι ε, μέρος της λύσεως και όχι του προβλήματος διότι το θέμα είναι να ξέρουμε τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιούμε τους κανόνες τους οποίους έχουμε διότι δεν χρησιμοποιούμε ε, πλέον το ευρωπαϊκό δίκαιο και το πιο απλό ίσως θα ήταν ε, να ε, κρατήσουμε μόνο τους νόμους τους οποίους θέλουμε να εφαρμόζουμε ή μπορούμε να εφαρμόζουμε. Θέλω όμως εδώ να αναφερθώ σε ορισμένες προτάσεις νομίζω ότι ε, βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο μεταξύ ε, ε, νομικής καταστάσεως και οικονομικής και πρέπει να δούμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Γι' αυτό είχε καταρτιστεί η έκθεση αυτή για τα προβλήματα του έκτου προγράμματος πλαισίου και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά αυτού του είδου διότι βλέπετε ότι διαφορετικά δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε Δηλαδή ε, θα πρέπει να υπάρχει μία πολύ κακή βαθμολόγηση και αν αντιληφθούμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά θα πρέπει να αλλάξουμε. Γι' αυτό καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα και ε, ε, είναι, δεν είναι πολύ εύκολο να εφαρμόσουμε το δίκαιο υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Γι' αυτό και θέλω να σας παρακαλέσω να μας πείτε και πάλι πώς απαντάτε συγκεκριμένο αυτό θέμα. Και μετά θα αναφερθώ και στο θέμα που έφυξε ο κύριος Λιμπεράσκη, δηλαδή τι μας αποδίδουν αυτά τα χρήματα, πού είναι τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας και πού αντικατοπτρίζονται, πού μπορούμε να τα διαβάσουμε, διότι χρηματοδοτούμε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε καν και μας κοστίζουν πάρα πολύ και δεν καταλήγουμε πουθενά. Άρα πολύ θα ήθελα να ξέρω αν τα αποτελέσματα αυτά τα διαθέτει μόνο η ερευνητική κοινότητα ή αν μπορούν να μεταδοθούν και στο ευρύ κοινό για να χαρεί. Είμαι μια εισηγήτρια στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και πιστεύω ότι θα έπρεπε την κατάσταση να μπορέσουμε να τη βελτιώσουμε και όχι να την επιδεινώσουμε. Είναι μια πρόκληση και τώρα υπάρχει συναπόφαση. Άρα είναι η κατάλληλη στιγμή ε, η Γενική Διεύθυνση Έρευνας ε, να εγκαταλείψει τους ε, κανόνες συμμετοχής διότι βλέπουμε ότι αυτοί είναι οι κανόνες που δημιουργούν πάντοτε τα προβλήματα τα υπόλοιπα θέματα τα έχουμε δρομολογήσει και μόνο οι κανόνες συμμετοχής μας δημιουργούν ακόμη προβλήματα. Ε, σε ποια ε, συμπεράσματα λοιπόν καταλήγεται σχετικά με το θέμα αυτό. Μήπως θα πρέπει να εγκαταλείψουμε ορισμένους κανόνες που εφαρμόζουμε ακόμη ε, κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να αντιληφθούμε πού καταλήγουμε με το, ε, με το δίκαιο διότι ε, θα ήθελα να ξέρω πού βρισκόμαστε και να μας πείτε πώς θα προχωρήσουμε. Όπως είπατε και στο τέλος, μας δώσατε πολλά θέματα τα οποία πρέπει να σκεφτούμε και συμφωνώ μαζί σας. Εγώ συγκεκριμένα έχω διαπιστώσει ε, πέντε θέματα τα, μέσα στα θέματα που θίξατε και όντως ε, η Επιτροπή αυτή δεν ήταν ποτέ μέρος του προβλήματος αλλά μάλλον συνέβαλε στην επίλυση και εγώ σας αντιμετωπίζω όπως και εσείς εμάς. Ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να εξετάσουμε είναι ότι αν θυμηθείτε τη συζήτησή μας πριν από τρία-τέσσερα χρόνια. Νομίζω ότι το πρόβλημα που έχουμε το δικαστήριο είναι ότι μιλάμε διαφορετική γλώσσα. Οι αριθμοί που φέρνουν, μάλλον το ελεκτικό συνέδριο, οι αριθμοί που φέρνουν ε, προσκομίζουν αυτοί και οι αριθμοί που έχουμε εμείς διαφέρουν και αυτό οφείλεται ε, στο ότι ε, δεν μιλούσαμε την ίδια γλώσσα ενώ διαμέσου των ετών μιλάμε πλέον την ίδια γλώσσα και πάμε πολύ καλύτερα. Όσον αφορά την απλοποίηση όπως πολύ σωστά είπατε θα υπάρξει μία ανακοίνωση εντός ενός δύο μηνών θα το έχετε μπροστά σας και όλα τα θέματα αυτά τα οποία εμείς εξετάζουμε ε, θα σας προσκομιστούν και θα, δούνε τι θα δείτε τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι... πώς προβλέπει να προχωρήσει όσον αφορά την ε, ε, αποπληρωμή. Βεβαίως το, το θα ήταν να μας δώσουν πίσω το 100% των ε, δαπανών. Αλλά έχει ε, εφαρμοστεί αυτό το σύστημα. Το 2008 όπως σας είπα καλύψαμε το 30% και το 2009 ε, πήραμε πίσω το 62%. Πάμε δηλαδή, είμαστε στο σωστό δρόμο και ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Για να είμαι ακριβής. Κάθε είδος κρίσεως, κατακρίσεως Δηλαδή ότι ε, έχει φτάσει η στιγμή να πληρώσει κανείς και η Επιτροπή να ανακτήσει τα ποσά που έδωσε είναι πολύ σωστή κριτική. Αυτό που ακούω εδώ είναι ότι πολύ σωστά μιλάτε, καταλαβαίνουμε την κριτική, θα κάνουμε καλύτερα του χρόνου, αλλά όσον αφορά την ε, κατάλληλη στιγμή για αποπληρωμή που ήταν πολύ κακή πριν από 2-3 χρόνια, τώρα τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ε, δεν είμαστε ακόμη στο επίπεδο που επιθυμούμε, αλλά έχουν γίνει μεγάλα βήματα προς τα μπρος όσον αφορά τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση. Ε, έχουμε ένα σύστημα, έχουμε αξιολογήσεις συχνές ε, και ε, έχουμε ήδη αξιολογήσει το πρόγραμμα πλαίσιο 7. Όλα δηλαδή τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί. Αλλά όταν μιλάμε για έρευνα θα πρέπει να καταλήγουμε στα αποτελέσματα ex τα οποία θα είναι στη διάθεση όλων. Αλλά για μια αξιολόγηση το βασικό θα πρέπει να υπάρχει εκ των προτέρων μια επιλογή. Δηλαδή από τις προτάσεις οι οποίες μας υποβάλλονται ή μάλλον υποβάλλονται στους ανεξάρτητους αξιολογητές, μία, από, μία στις πέντε επιλέγονται. Οι τέσσερις πετιούνται και ελπίζουμε ότι για την αξιολόγηση έχει ληφθεί η σωστή γιατί οι κύριοι αυτοί είναι, είναι επαγγελματίες και ε, αν υπάρχει μία κατάκριση κάναμε μία ανάλυση και περίπου το 90% των αξιολογητών είπαν ότι η διαδικασία που διαπιστώνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον, είναι, ε, τουλάχιστον αντικατοπτρίζει την κατάσταση των κρατών μελών ή και ακόμη περισσότερο. Οπότε δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω αυτή τη διαδικασία επιλογής. Ξεχνάμε πολλές φορές ότι πρόκειται για πολύ σημαντικά παράθυρα μέχρι, μέσω των οποίων ε, εξετάζουμε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, ε, για ε, το τρέχον έτος ε, δεν ξέρω αν θα έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Σε 10 χρόνια ή σε 20 είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να παράγουμε ε, βραβεία Νόμπελ. Αλλά ίσως τώρα μπορεί να ακόμη να χρηματοδοτούμε 10-20% προγραμμάτων τα οποία είναι τελείως λάθος και δεν θα αποδώσουν καθόλου. Ατυχώς είναι μέσα στο σύστημα. Επίσης ένα μέλος της Επιτροπής σας ε, έθεσε μία ερώτηση ότι χρειάζεται μία δημοσιονομική αναθεώρηση και συμφωνώ ότι επιβάλλεται διότι διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να είσαστε ε, βέβαιοι ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το προχωρήσω ακόμη και αν έχω λίγα χρόνια πίσω μου και όχι πολλά. Η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που επανέρχομαι σε αυτό το θέμα και πάλι. Όσον αφορά την ε, ε, ε, μη χρήση των πόρων είναι ένα θέμα που μας δημιουργεί προβλήματα διότι δεν τα βγάζουμε πέρα και γι' αυτό αρνούμαστε την απαλλαγή καμιά φορά. Σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται με τους γεωργούς. Στους γεωργούς δεν θα σκεφτείτε σκεφτόμασταν να αρνηθούμε κάτι. Θέλουμε να ελέγχουμε τουλάχιστον 5%. Ε, ενώ ε, εδώ ξεκινήσαμε με 1% και επικοιτάμε να φτάσουμε στο 5%. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει από πολύ χαμηλά. Και εγώ σαν εκλεγμένη να έχω πρόβλημα. Πέστε μου τι πρέπει ε, να πω στη συνάντηση που θα έχω το επόμενο Σάββατο. Ε, τι μπορώ να τους πω. Ελπίζω να μην ξέρουν. Αλλά αν με ρωτήσουν γιατί ε, τους γεωργούς τους αντιμετωπίζουμε διαφορετικά από την έρευνα όσον αφορά τις επαληθεύσεις, πέστε μου τι πρέπει να τους απαντήσω. Το γεωργικό σύστημα δεν το κατέχω ιδιαίτερα. Αλλά σας πιστεύω. Νομίζω ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε εδώ είναι πρώτον να έχουμε μια αυστηρή διαδικασία επιλογής. Επιλέγεται ένα στα πέντε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αγγίηση αυτή τη στιγμή ότι τα μέτρα εξάντε εκ των προτέρων θα μας απαλλάξουν από όλα τα σφάλματα στο σύστημα, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε έναν εκτενή έλεγχο εκ των υστέρων. Τώρα πόσο εκτενεί δεν ξέρω. Αν θέλουμε να απαλλαγούμε από το σύστημα αυτό και συμφωνώ με αυτό που είπατε, το σύστημα αυτό κατά πάσα πιθανότητα από τη φύση του οδηγεί σε λάθη. Άρα πρέπει να πάμε προς την κατεύθυνση την οποία και εσείς επισημάνατε. Δηλαδή μέση όρη, καταποκοπή ποσά. Αλλά εδώ στην περίπτωση αυτή υπάρχουν άλλα προβλήματα. Εγώ προσπάθησα να τα καλύψω όλα τα θέματα όσο μπορούσα αυξήσουμε τον αριθμό των ελέγχων. Αλλά αν θέλετε την ειλικρινή μου άποψη, η σωστή κατεύθυνση δεν είναι αυτή. Γιατί τελικά μπορούμε να ελέγχουμε το 100% αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα για την έρευνα στην περίπτωση αυτή. Κύριε Επίτροπε, με ενδιαφέρουν τα πιστοποιητικά ελέγχου, τα οποία διαβάσαμε. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την αξιολόγηση αυτών των πιστοποιητικών αξιολογήσεως. Θεωρείτε ότι το σύστημα είναι λογικό και αν όχι τι εναλλακτική λύση θα προτείνατε και μία συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με το ανώτατο όριο το ανώτατο των 375.000 ε, για ε, ε, προγράμματα ερεύνης για τα οποία καταρτίζεται ένα πιστοποιητικό αξιολογήσεως Πώς καταλήγουμε σε αυτό το ποσό. Ε, υπάρχει κάποιο επιχείρημα. Ε, μπορείτε να μου πείτε για ποιο λόγο έχει επιλεγεί αυτός ο αριθμός και όχι κάποιος άλλος. Και τέλος ποιο είναι το ποσοστό των προγραμμάτων που είναι κάτω από το ανώτατο επίπεδο των 375.000 ευρώ και τι γίνεται με τους ελέγχους σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρώτο, το σύστημα των πιστοποιητικών ελέγχου έδωσε ένα αποτέλεσμα, λιγότερα σφάλματα πριν, από ότι πριν εισαχθεί το σύστημα. Ωστόσο, αν μιλάμε για το FP6, το πλαίσιο 6, όπου δεν υπήρχε κατόφλι, που υπήρχαν αιτήματα δικαιολογημένα τα πράγματα ήταν αρκετά πολύπλοκα και το κόστος ψηλό. Γι' αυτό ε, εισηγάγαμε το 375.000 όριο. Έγινε μια προσωμείωση με μοντέλο 5% απόκληση όπως μου εξηγούν οι συνεργάτες μου γιατί για να σας πω την αλήθεια δεν το ήξερα αυτό πριν Έχουμε και εμεί εμπειρογνώμονε. Μπορείτε και εσεί να ζητήσετε από κάποιο εμπειρογνώμονε να σα το εξηγήσει. Δεν είναι αυθαίρετα τα νούμερα. σω το 5% να είναι αυθαίρετο, αλλά με βάση το 5% από εκεί και πέρα ο υπολογισμό είναι πολύ συγκεκριμένο. Πρόεδρο. Ευχαριστούμε. Δευτερολογεί ο κ. Βουλευτή. Κύριε Πίτροπε, δεν μου απαντήσατε πόσο ποσοστό των ερευνητικών προγραμμάτων είναι κάτω από αυτό το ανώτατο όριο των 375.000 ευρώ. Δεν γνωρίζω. Θα σας απαντήσω γραπτός ή αν κάποιος σου το γνωρίζει από το επιτελείο μου, αλλά νομίζω γραπτός θα σας απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, λέει ο κύριο Στάς, για τη συνεργασία μας τα τελευταία πέντε χρόνια. Κάθε φορά που υπήρχαν προβλήματα από την πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου, εσείς δράσατε προδραστικά. Ήρθατε στο κοινοβούλιο, συζητήσατε με τους συναδέλφους μας. Σωστό αυτό. Καλό παράδειγμα. Μία μικρή ερώτηση. Μας είπατε ότι όταν κάποιος ζητάει επιστροφή για την έρευνα, όταν ζητάτε μάλλον επιστροφή, το 40% του ποσού αυτού δεν επιστρέφεται. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αρνούνται να συνεργαστούν όταν τους ζητάτε να επιστραφούν τα χρήματα αυτά, γιατί το 40% των φορέων σημαίνει ότι είναι πολλοί. Είναι πάντα οι ίδιοι που κάνουν αυτά τα πράγματα είναι στους ίδιους τομείς έρευνας. Πρόκειται για πανεπιστήμια, ερευνητικά Ινστιτούτα. Μπορείτε να μας πείτε κάτι. Απάντηση. Είναι πολύπλοκο το σύστημα. Πρέπει να, να ξεκαθαρίζουμε τις, την ανάκτηση ποσών και τις, τα πρόστιμα, η κυρώσεις. Η ανάκτηση ποσών, recoveries, είναι όταν με έναν έλεγχο διαπιστώνουμε ότι έγινε ένα σφάλμα και το διορθώνουμε. Είτε ζητάμε τα λεφτά ή αφαιρούμε τα χρήματα αυτά από μελλοντικές πληρωμές. Είπα ότι σιγά σιγά εισάγουμε ένα νέο σύστημα. Το, το σύστημα αυτό μάλλον. Το 2008 είχαμε το 30% ανάκτησης αυτό που είχαμε εντοπίσει. Τώρα ανεβαίνουμε σε ποσοστό. Πρέπει πρώτα να γίνει ο εντοπισμό και μετά να γίνει η ανάκτηση. Πάντα υπάρχει μια χρονική υστέρηση. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Πρέπει να βελτιωθούμε, αλλά η ψαλίδα κλείνει. Άλλο πράγμα τώρα είναι η ανάκτηση ποσών που στηρίζονται σε χρονική προβολή προς το μάλλον. Δηλαδή, εντοπίζουμε ένα συστημικό σφάλμα, κάνουμε προβολή στο μέλλον, αλλά βέβαια τα πράγματα είναι λίγο πιο λεπτά. Δηλαδή, έχουμε πολλές καταγγελίες και παράπονα και η δική σας επιτροπή μας ζήτησε να κάνουμε κάτι. Με βάση όλα αυτά, ε, εγκρίναμε αυτή την πρόσφατη ανακοίνωση του Δεκεμβρίου για να λυθεί το θέμα αυτό σωστά. Δεν είναι ότι δεν θα γίνουν οι ανακτήσεις. Θέλουμε να απλουστεύσουμε το σύστημα με τον ε, καταποκοπή συντελεστή. Και μερικές από αυτές τις δηλώσεις για το κόστος έγιναν καλοπροαίρετα. Γιατί εσωτερικά αυτό το σύστημα εφαρμοζόταν σε ορισμένες χώρες. Τώρα, για το μέλλον, λέμε οι κανόνες θα πρέπει να τηρούνται 100%. Ας την πούμε αυτή η μεταβατική μέθοδο. Βάζουμε περισσότερη τάξη. Βέβαια, αν εμείνουμε στο μοντέλο κόστους που έχουμε σήμερα και στο μέλλον. Το πρόβλημα που το αναγνώρισαν και άλλοι, το τόνιστε δηλαδή το συνέδριο, είναι οι κυρώσεις β' πρόστιμα. Στο FP, ε, πρόγραμμα πλαίσιο 7, είμαστε υποχρεωμένοι να γίνει αυτή η ανάκτηση, ενώ στο 6 δεν προβλεπόταν αυτό. Υπάρχουν δύο είδη κυρώσεων. Η μία είναι οι οικονομικές ε, ποινές και άλλη είναι κάπως διαφορετικό. Στην έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου αναφέρεται. Σας πληροφορώ ότι το 2009 αρχίσαμε τις ανακτήσεις από τα πρόστιμα, ζητάμε πίσω τα χρήματα, έτσι ώστε το 2009 αυτό ίσχυσε αυτή η έννοια για το 30% τις ε, τα πρόστιμα δεν το ξεκινήσαμε ακόμα γιατί χρειάζεται απόφαση της Επιτροπής και ο Γενικός Διευθυντής μελετάει το θέμα αυτό. Χρειάζεται μια λύση μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2010 για τα πρόστιμα και θα ισχύσει αυτό για το πρόγραμμα πλαίσιο 6. Για το πρόγραμμα πλαίσιο 7 σας είπα η κατάσταση είναι διαφορετική. Παναλαμβάνω είναι περίπλοκη η κατάσταση. Ωστόσο ε, νομίζω ότι σας έδωσα στοιχεία για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Πρόεδρος, μας έχουν μείνει τρία-τέσσερα λεπτά. Δύο-τρεις συνάδελφοι, παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι. Πρώτον, ο κύριος Νόακ από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον παρακαλώ ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να προσθέσω ε, στην ερώτηση προς τον, ε, ή στην ερώτηση μάλλον του κυρίου Λιμπεράτσκη, του Επιτρόπου, αν θα έπρεπε να αλλάξουμε το σύστημα για τη δαπάνη για την έρευνα και για τη χρηματοδότηση για την έρευνα. Όχι είναι η απάντηση. Χρειαζόμαστε ένα μείγμα εργαλείων και μέσων προς όφελος των δικαιούχων, των αναγκών τους, των οργανώσεων, των οργανισμών που μπορεί να είναι υποκοπή ποσό αλλά μπορεί να είναι και μια κατάσταση βεβαιωμένου κόστους Όσο πιο διαφοροποιημένη η λύση, όσο πιο καλό το μείγμα, στο το πούμε αυτό, το, αυτή η σύνθεση των εργαλείων, τόσο πιο καλή. Αυτή, αυτά λέει η σύστασή μας. Πρόεδρος, η, ο Επίτροπος νομίζω θέλει να προσθέσει κάτι. Μάλιστα, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Δόκτωρ Νόακ του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πρόθεσή μου δεν ήταν να πω ας κάνουμε επανάσταση. Μερικές αλλαγές θέλουμε. Στα προγράμματα πλαίσιο 6, 7 και 8 δεν είναι δυνατόν να εισαχθούν αυτές οι αλλαγές. Το αν είναι πιο ουσιώδεις αλλαγές, είναι, ναι, συμφωνώ. Αλλά γι' αυτό η πρότασή μου και εμένα είναι ένα μείγμα ανεκτού κινδύνου λάθους και απλοποίηση. Πρόεδρος, ο κύριος Βόγκαν, σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, την περασμένη εβδομάδα η, Πρόεδρος, η Επίτροπος ε, μίλησε για τις προθέσεις της σχέση με το, ε, με το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Είπε ταυτόχρονα ότι το σύστημα θα πρέπει να απλοποιηθεί. Και αυτό το ακούσαμε και από σας σήμερα. Αυτό το οποίο δεν βλέπω όμως πάντα είναι κάποιο πρακτικό παράδειγμα ε, του τι θα πετύχουμε με τον τρόπο αυτό. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκα με τα πανεπιστήμια στην Ουαλία και όλοι μιλούσαν για το ίδιο πράγμα. Απλοποίηση ε, του προγράμματος PFP. Ε, παράδειγμα που μας έδωσαν. Πρώτα απ' όλα μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο όταν γίνει η προκήρυξη, καταλαβαίνετε εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδυαστούν τα σχέδια και δεύτερον μπορούν να συνδυαστούν τα σχέδια μόνο αν υπάρχουν εταίροι και από άλλα κράτη-μέλη, το οποίο περιπλέκει πολύ περισσότερο τα πράγματα. Έχετε εξετάσει κάποια από τα στοιχεία αυτά και θα ενθαρρύνετε την Επίτροπο να τα δει τα στοιχεία αυτά και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Ναι, η απάντηση είναι οποιαδήποτε δυνατότητα ε, προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να εξεταστεί. Αλλά κοιτάξτε, εγώ έχω απελπιστεί, δεν πιστεύω πια ότι θα υπάρξουν παράπονα από τους χρήστε ότι θα μπορούμε να τα εξαλείψουμε. Ευχαριστούμε. Τελευταία ερώτηση, κυρία Γκρέσλε, πάρα πολύ σύντομα. Όσον αφορά τις γραπτές απαντήσεις, θέλω δύο νούμερα. Πρώτον, όσον αφορά τους ελέγχους ex post, το ποσοστό τους, και ε, ε, των ετοιμάτων που οδήγησαν σε ε, επιτυχία. Ευχαριστώ. Θέλω αυτά τα δύο νούμερα. Το μόνο που μπορώ να σα υποσχεθώ είναι ότι θα τα πάρετε γραπτά. Ναι, γιατί ε, ότι, βεβαίω όταν μιλάμε για τι λεπτομέρειε καλύτερα να είμαστε σίγουροι και να τα στέλνουμε γραπτά. Σα ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για το γεγονό ότι ήρθατε εδώ σήμερα. Και τώρα να περάσουμε στην δεύτερη ακρόαση με τον Επίτροπο Αντώνιο Ταγιάννη. Α, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν ο εκπρόσωπο του συνεδρίου θέλει να προσθέσει κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία είπαμε πριν από λίγο ε, προ τον Επίτροπο το ε, υπεύθυνο για τι μεταφορέ. Ίσχυουν αυτά τα οποία είπατε και πριν από λίγο. Κύριε Νόκα, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, νομίζω ότι με την εισαγωγική μου, με την εισαγωγή μου κάλυψα όλα τα σημεία. Είπα ό,τι ήθελα να πω. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα, αλλά δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Ωραία. Νομίζω τώρα μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον ε, εισηγητή, στον κύριο Λιμπεράσκη, για να μπορέσει να μας παρουσιάσετε τα ζητήματα. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ξεκινήσω ναι. με την εξή ερώτηση όσον αφορά το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Ξέρουμε ε, ότι έχει ξεπεράσει ε, κατά πολύ τον προπολογισμό του, τη διάρκεια του και βεβαίως ε, το συνέδριο ήδη έχει εκφράσει την άποψή του. Κύριε Αντιπρόεδρε, τι συνέβη με το Γαλιλαίο και τι προοπτικές έχουμε. Πόσο θα κοστίσει σε τελευταία ανάλυση και πότε θα έχει ολοκληρωθεί. Ποια είναι η άποψή σας Βεβαίω, ε, εσεί αλλάζετε αρμοδιότητε στο μέλλον. Αλλά θα ήθελα να ακούσουμε τις, ε, αυτά τα οποία έχετε να μα πείτε. Επίτροπε, αν θέλετε. Βέβαια, ε, δεν ξέρω, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι σχέση με το ελεκτικό συνέδριο, να απαντήσετε απευθεία στον εισηγητή. Ναι, καλησπέρα σα. αν συμφωνείτε, θα ήθελα να κάνω μία σύντομη εισαγωγική παρουσίαση. Εκεί όπου θα μιλήσω και για τον Καλλιλέο Και στη συνέχεια θα ε, επισέλθω σε ερωτήσει, να απαντήσω. Έτσι για να πάρετε μία συνολική εικόνα ε, όλων αυτών που αφορούν τι δικέ μου αρμοδιότητε ε, ε, τώρα στο τέλο τη θητεία μου. Και απαντώ απευθεία στον εισηγητή θα εξακολουθήσω να ασχολούμαι με τον Γαλιλαίο ε, εάν ε, εγκρίνει τη νέα επιτροπή και με τις νέες μου Είναι ένα θέμα το οποίο θα εξακολουθήσω να το παρακολουθώ και τα επόμενα πέντε χρόνια και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε για να μιλήσουμε και για τον Γαλιλαίο. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Σιγητά, ε, ε, κύριε Νόακ, κυρία Καλουλάιτ, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν το συγκρίνουμε με τα 7 δις ε, ευρώ ε, της έρευνας του 2008, καταλαβαίνω ότι οι δαπάνες για τις μεταφορές που μόλις ξεπερνούν το 1 δις ευρώ μπορεί να φαίνονται ελάχιστες. Αλλά δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Πάντως καταλαβαίνω πολύ καλά το λόγο για τον οποίο προσκαλέσατε σήμερα εδώ. Και με μεγάλη μου ευχαρίστηση βρίσκομαι σήμερα ενώπιον της Επιτροπής σας για να σας πω τι κάναμε και να απαντήσω και στις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, 1 δις ευρώ από αποτελούν ένα σημαντικό ε, χρηματικό ποσό, ιδιαίτερα μέσα στο σημερινό ε, οικονομικό ε, περιβάλλον όσον αφορά τον προπολογισμό και την απασχόληση. Και δεύτερον, γιατί τα βασικά προγράμματα ε, ε, τα οποία αφορούν ε, το, Γαλλιό για παράδειγμα και τα διευρωπαϊκά δίκτυα είναι σχέδια εχμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να αποτελέσουν υπόλοιπη. Έτσι, βεβαίω είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να μειώσουμε το περιθώριο σφάλματος και με αυτή την έννοια χαίρομαι ιδιαίτερα και συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο κ. Ποτότσινικ και όσον αφορά την απλοποίηση ε, τη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και όσον αφορά το επίπεδο ε, κινδύνου. Είμαι ικανοποιημένο λοιπόν γιατί η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για το 2008 δεν έδειξε όσον αφορά αυτά τα σημαντικά σχέδια κανένα νέο στοιχείο το οποίο ε, δεν έχει ληφθεί υπόψη ή δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο διαχείριση από την Επιτροπή. Σε γενικέ γραμμέ πρέπει να πω ότι το μήνυμα του συνεδρίου κατά την άποψή μου είναι θετικό. Όσον αφορά τι μεταφορέ απαραδείχεται μόνο ένα σφάλμα μη συστηματική φύσεω που αφορά το σχέδιο ε, για τα ευρωπαϊκά TNT ε, Λιόν Τωρίνο το οποίο αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να διορθώσουμε όσον αφορά την έρευνα που συνδέεται με τι μεταφορέ, θέμα το οποίο συνδέεται και με την προηγούμενη συζήτηση με τον συνάδελφο Τότσινγκ θέλω να πω το εξή. Πρώτον, ότι όσον αφορά την έρευνα που αφορά τι μεταφορέ, εδώ το τμήμα τη έρευνα που συνδέεται με τι ε, μεταφορέ καλύπτει ένα, σχετικά χαμηλό ποσοστό τη συνολική, του συνολικού προπολογισμού για την έρευνα, 0,2 δι, επί συνολικού ποσού 6,7 δι. Δεύτερον, το ποσοστό τη έρευνα το οποίο συνδέεται με τι μεταφορέ συμβάλλει στο να μειώσει το μέσο όρο ε, του ε, ποσοστού των όπω εντοπίστηκαν από το ε, συνέδριο ε, στο σύνολο του τομέα τη έρευνα. Αλλά δεν θέλω αυτή τη στιγμή να σα πω ότι επαναπαυόμαστε στι δάφνε μα. Ε, το αντίθετο. Όλοι μα εργαζόμαστε εντατικά για να μειώσουμε περαιτέρω το ποσοστό του σφάλματο, ακολουθώντα το τελικό στόχο του να λάβουμε μία αξιολόγηση από το συνέδριο χωρί σφάλματα. Στο, στο, όσον αφορά το θέμα αυτό, από την αρχή του 2008, δηλαδή έξι μήνε πριν από τη δική μου ανάληψη των καθηκόντων ε, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ως Επιτρόπου υπεύθυνου για, την, ε, για τις μεταφορές, η Γενική Διεύθυνση Τρέν επέβαλε σημαντικέ και ριζικέ αλλαγέ όσον αφορά τον τρόπο χρηματοδότηση. Και σίγουρα αυτή η προσπάθεια συνεχίσει και στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία εντάσσονται και στι απαντήσει που αποστήλαμε πριν από την σημερινή ακρόαση. Πριν ε, ε, τελειώσω την εισαγωγή μου και απαντήσω στην πρώτη σας ερώτηση που αφορά το Γαλιλαίο, θα ήθελα να σταθούμε για λίγο σε αυτό το σχέδιο, το οποίο εντάσσεται και στις ε, σημερινές μου αρμοδιότητες και που ε, χάρισε στη δική σας υποστήριξη. Είναι λοιπόν και θέμα το οποίο θα με απασχολήσει... στην προσοχή μου θετία. Το 2008, που είναι έτος αναφοράς κύριε Πρόεδρε για τη σημερινή συζήτηση, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά το ε, παγκόσμιο σύστημα πλοήγησης, δορυφορικής πλοήγησης. Το 2008 αναδιαρθρώθηκε ριζικά, διότι μέχρι το τέλος του 2007 είχε να αντιμετωπίσει πολυάριθμες προκλήσεις. Προκλήσεις που διευκρινίστηκαν συγκεκριμένα και μέσα στην ειδική έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου που αφορά τη διαχείριση του προγράμματος στο χρονικό διάστημα 2003-2006. Είμαι πεπισμένος ότι σήμερα η ριζική αναδιάρθρωση του προγράμματος του 2008 αρχίζει αυτή τη στιγμή να μα οδηγεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα θετικά κατά την άποψή μου. Όταν το συνέδριο θα εξετάσει εκ νέου το πρόγραμμα, είμαι σίγουρο ότι θα εντοπίσει σημαντικέ ε, βελτιώσει όσον αφορά τη διαχείριση ενό προγράμματο που πάνω απ' όλα είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο και καινοτόμο. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι στι 7 Ιανουαρίου 2010, αφού ενημερώθηκε ε, το ε, διοργανικό η Διοργανική Επιτροπή Γαλιλαίο, Διοργανικό Πάνελ Γαλιλαίο, ανακύρωσα, ε, ανακοίνωσε συγγνώμη, την προκήρυξη τριών σημαντικών διαγωνισμών ε, για την, ε, που αφορούν την, την επιχειρησιακή ικανότητα του Γαλιλαίου. Ε, οι αποφάσει ε, αυτέ ε, αφορούν τη Σύμβαση για τι υπηρεσίε υποστήριξη του συστήματο, τη Σύμβαση για την πρώτη παρτίδα 14 δορυφόρων και, και μια πρώτη σύμβαση για την εκτόξευση των 10 δορυφόρων. Όσον αφορά την πρώτη παρτίδα 14 δορυφόρων, μιλάμε για ένα συνολικό ποσό 566 εκατομμύρια ευρώ και επελέγει η εταιρεία OHB System AG, γερμανική επιχείρηση. Ε, που έχει και ε, θηγατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι υπηρεσίε υποστήριξη του συστήματο ανατέθηκαν στην ε, Tails Alinea Space, Ιταλική εταιρεία. Η σύμβαση αφορά το ένα ποσό 85 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, Διαστημικού Οργανισμού για την ενσωμάτωση και την επαλήθευση του συστήματος Γαλιλαίου. Η σύμβαση για τι υπηρεσίε εκτόξευση ανατέθηκαν στο Ariane Space, γαλλική επιχείρηση, για συνολικό ποσό 397 εκατομμύρια ευρώ για πέντε εκτοξεύσεις Σογιούς. Θα ήθελα επίση να επαναλάβω ότι εμεί, και, όταν και, και αυτό το εμεί σημαίνει Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματο, καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για να εγγυηθούμε ότι όλα αυτά θα γίνουν με ιδιαίτερα ισότιμο και διαφανή τρόπο και τα αποτελέσματα ε, θα εκφράζουν την καλύτερη σχέση ποιότητα-τιμή. Δεύτερον, θέλω να τονίσω ιδιαίτερα τη σημασία αυτή τη ανακοίνωση. Πράγματι, μετά από 18 μήνε, κατά τη διάρκεια των οποίων συγκεντρώσαμε την προσοχή μα στη διαδικασία δημοπράτηση, αρχίζουμε τώρα τη μετάβαση προ την φάση εφαρμογή του συστήματο Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκής ε, δορυφορικής πλοήγησης. Με την ε, ανάθεση των ε, συμβάσεων που ανακοινώθησαν, μπορούμε τώρα να καθορίσουμε πιο συγκεκριμένα τον προγραμματισμό του Γαλιλαίου και να προγραμματίσουμε καλύτερα και τις δημοσιονομικές ανάγκες. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα γιατί μπορώ να σα ανακοινώσω ότι ε, ε, τώρα ε, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για να δώσουμε στου πολίτε, στου Ευρωπαίου πολίτε, τι πρώτε υπηρεσίε πλοήγηση από τι αρχέ του 2014. Άλλε τρει παρτίδε που αφορούν τη διαδικασία δημοπράτηση του Γαλιλαίου βρίσκονται ακόμα στη φάση αξιολόγηση. Αφορούν τι χερσαίε υποδομέ, χερσαίε υποδομέ για τι αποστολέ και για τον έλεγχο, καθώ επίση τι επιχειρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία ανάθεση αυτών των συμβάσεων το πολύ μέχρι ε, το ίμιση του 2010. Στη συνέχεια θα ανατεθούν οι συμβάσει για την κατασκευή και την εκτόξευση των υπολείπων ε, δορυφόρων με στόχο να έχουμε φτάσει στην πλήρη ε, επιχειρησιακή ικανότητα που στηρίζεται σε 30 δορυφόρου. Αυτό τι σημαίνει συνοπτικά. Στο τέλο αυτού του έτου προβλέπεται η εκτόξευση σε τροχιά των πρώτων δύο ε, λειτουργικών δορυφόρων. Το 2011 θα ακολουθήσουν άλλοι δύο και μέσα στο τρίτο ε, τρίμηνο του 2012 θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την εκτόξευση ενό ζεύγου δορυφόρων κάθε τρει μήνες. Οι ανοιχτέ υπηρεσίε Open Service οι ρυθμιζόμενε δημόσιε υπηρεσίε, public regulated service και οι υπηρεσίε έρευνα και διάσωση, search and rescue service, θα είναι λειτουργικέ από τι αρχέ του 2014. η πειραματική φάση τη υπηρεσία για τη διάσωση των ανθρώπων, safety of life service και τη εμπορική υπηρεσία, commercial service, θα ξεκινήσουμε στο 2014 και οι υπηρεσίε ε, θα δοθούν μόλι το Γαλιλαίο ε, φτάσει στην πλήρη του επιχειρησιακή ικανότητα, όπω σα είπα, με αυτού του 30 δορυφόρου. Όπω βλέπετε λοιπόν, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον Γαλιλαίο. Τώρα, ε, ο εισηγητή ε, ε, στη συζήτηση αυτή θέτει το εξή πρόβλημα. Μα υπάρχουν αρκετά χρήματα και γιατί υπάρχει αυτό ο κίνδυνο περαιτέρω αύξηση των προβλέψεων. Γιατί αναφέρθηκε στον τύπο η αύξηση των δαπανών για την ολοκλήρωση αυτού του φιλόδοξου ευρωπαϊκού προγράμματο. Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί και για, και για λόγου υποστήριξη βιομηχανία, αλλά και για πολιτικού λόγου επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω ξέρετε, υπάρχει το αμερικάνικο σύστημα, το GPS, υπάρχει το ρωσικό, υπάρχει το, το, το σύστημα των Κινέζων, ε, τη Ινδία, ε, όλα αυτά τα συστήματα τα οποία βρίσκονται στη φάση τη αναδίπλωση. Εδώ μιλάμε λοιπόν για ένα ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο ε, θα γίνει παγκόσμιο ο πατέρα του Γαλιλαίου, το έγκνο, το οποίο ήδη λειτουργεί, όπω γνωρίζετε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά μόνο την Ευρώπη είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ενώ τον Γαλιλαίο, ε, το οποίο ε, αποτέλεσε αντικείμενο πλήρου χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την αρχική αλλαγή, θα θυμάστε, ε, όπου ήταν σύμπραξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα, τώρα έγινε κοινοτικό πρόγραμμα. Θα ξέρετε πολύ καλά τα, τα γεγονότα και πώ εξελίχθησαν. Δεν χρειάζεται να τα υπενθυμίσω. Αυτή η αλλαγή οδήγησε και σε ε, διαφορετική οικονομική ε, ανάληψη υποχρεώσεων ε, και διαφορετική χρησιμοποίηση κονδυλίων. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθο. Τώρα, εμεί τη διαχείριση της έρευνας και των δημοπρατήσεων το έχουμε αναθέσει στον Ευρωπαϊκό, στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση Διαστήματος παρόλο που η τελική απόφαση ανήκει σε εμά. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι το καλό. Ε, γιατί ε, με αυτόν τον τρόπο συνδυάζουμε ε, την άριστη συνεργασία με το καλό αποτέλεσμα. Τώρα, το οικονομικό πρόβλημα ποιο είναι. Σήμερα, με τις αποφάσεις που λάβαμε, δηλαδή όλη η εργασία που μπορούμε να κάνουμε μέχρι το 2014, που θα έχουμε την έναρξη της, επιχειρησιακή της, της επιχειρησιακής φάσης του Γαλιλαίου, θα είμαστε απόλυτα λοιπόν μέχρι στον προκαθορισμένο προπολογισμό μέχρι τότε βρισκόμαστε γύρω στα 3,6 δις ευρώ. Εκεί είναι. Αλλά έχουμε αυξήσει κυρίω όσον αφορά τα συστήματα εκτόξευσης. Ε, η άνοδος των τιμών τη αγοράς όσον αφορά τα συστήματα εκτόξευσης αυξήθηκε από 60% 80%. Εμείς, ε, όπως είπα ε, και στην ε, εισαγωγική μου παρουσίαση, προσπαθήσαμε μέσα από τη διαδικασία δημοπράτησης ε, να ε, σεβαστούμε ε, απόλυτα τα ανώτατα όρια τα οποία έχουν προκαθοριστεί. Άρα, αν θέλετε, ε, ε, σεβαστήκαμε με τον καλύτερο τρόπο κατά την άποψή μου και τον πιο αποτελεσματικό τη σχέση ποιότητα-τιμή ε, έτσι ώστε να προσπίσουμε τα συμφέροντα των πολιτών. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση, Πρόεδρε, αν μιλάμε για την συνολική υλοποίηση του προγράμματος Γαλιλαίο και κατά πόσο θα απαιτηθούν περαιτέρω κονδύλια πέραν αυτών που ήδη έχουμε προβλέψει, να σας πω και το είπα και κατά την ακρόαση ως ε, επίτροπος που θα εξακολουθήσω να έχω ε, την ε, ευθύνη για τον Καλλιλέο, παρόλο που θα γίνει από μια άλλη σκοπιά, από την έρευνα, από τη βιομηχανία, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν θα υπάρξουν συμπληρωματικό κόστος. Δεν θα υπάρξει συμπληρωματικό κόστος. Αυτό το αποκλείουμε. Αλλά εάν υπάρξει τέτοια ανάγκη, πρέπει να δούμε τα εξή. Πρώτα απ' όλα να δούμε για ποια αύξηση μιλάμε αφού το καθορίσουμε, θα έρθω στο Κοινοβούλιο για να σε ενημερώσω, γιατί αυτό αποτελούσε πρακτική μου και στο παρελθόν. Και νομίζω ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά και με τη διοργανική ε, ομάδα εργασία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος, ε, κάποιο μέλο του Κοινοβουλίου που εργάζεται και σε αυτή την ομάδα. Α, έχουμε την κυρία Νίμπλερ. Ε, με, ήταν η πριν η κυρία Νίμπλερ με τη διοργανική ομάδα. Θα δούμε λοιπόν εάν θα πρέπει αν για να ολοκληρώσουμε το, το Γαλιλαίο απαιτηθούν περαιτέρω χρήματα, σα το λέω, θα έρθω αμέσω να σα ενημερώσω για τυχόν τέτοιε ανάγκε. Και βεβαίω και το Συμβούλιο ε, που είναι ε, το, το άλλο σκέλο τη διοργανική ε, ομάδα, έτσι ώστε να ληφθεί μια απόφαση στα πλαίσια τη μέγιστη διαφάνεια. Νομίζω ότι όσον αφορά το θέμα αυτό, πρόκειται για χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Πρόκειται για ένα κοινοτικό πρόγραμμα, ευρωπαϊκό πρόγραμμα μεγάλη εμβέλεια, για μεγάλη πρόκληση. Και το υπενθυμίζω. Εδώ ε, βεβαίω τα χρήματα είναι πολλά, αλλά αν κάνουμε του λογαριασμού. Και το έκαναν ορισμένε ε, άλλε εταιρείε για το πόσα χρήματα θα εξοικονομήσει η Ευρώπη. Όταν αρχίσει να λειτουργεί το Γαλιλαίο, νομίζω ότι μέσα σε 10-15 χρόνια θα εξοικονομήσουμε 90 δις ευρώ. 2,6 λοιπόν δις ευρώ επενδύουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, βεβαίως. Μπορεί να απαιτηθούν και συμπληρωματικέ επενδύσει, εάν θέλουμε να ολοκληρώσουμε το σύστημα και προκύψουν άλλε ανάγκε. Μετά τη θέση σε λειτουργία του 2014, και το ξαναλέω, μέχρι το 2014 θα αρχίσει να λειτουργεί το Γαλιλαίο ε, από λειτουργική άποψη. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτόξευση όλων των δορυφόρων και η θέση σε λειτουργία του. Εάν θέλουμε να φτάσουμε στου 30 δορυφόρου κτλ., θα δούμε εκεί κατά πόσο να απαιτηθούν ε, και παραπάνω χρήματα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε και η δήλωσή σας ε, και τα ε, ε, θέματα που θίξατε είναι πολύ εντυπωσιακά όπως είναι και τα επιτεύγματά σας σε αυτό το τομέα. Εάν λοιπόν η Επιτροπή αυτή αποφασίσει να να παραμείνετε εις το, εις το χαρτοφυλάκιο αυτό προς το παρόν προβλέπει ο κύριος Κάλλας. Ε, όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Για κάθε χρόνο παραπονιόμαστε ότι τα χρήματα που διατίθενται για αυτά τα προγράμματα είναι εν τρίτον, εν τέταρτο του ποσού που έχουμε ζητήσει και ε, αναμένουμε. Έχετε προβλέψει δέκα νέα ε, γραφεία. Κύριε Επίτροπε, ποιο είναι το αποτέλεσμα, τι κόστισες και είσαστε ικανοποιημένος από το κόστος και τα αποτελέσματα αυτών των γραφείων. Οικονομικά το σύστημα αυτών των γραφείων είναι διάφανο για σας. Ευχαριστούμε. Επίτροπε. Εκτός μικροφώνου. Μάλιστα, όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα, εμεί θα πρέπει να αξιολογήσουμε το ζήτημα από πολιτική άποψη και τη τελευταία να να, η αξιολόγησή μα αυτή είναι θετική. Οι χρηματοδοτήσει που επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και κοιτάξτε, εγώ υπέγραψα μία σειρά από εγκρίσει για χρηματοδοτήσεις τα Χριστούγεννα του 2008 για μια σειρά από πολύ σημαντικά προγράμματα. Λοιπόν, ε, ε, ε, πραγματικά νομίζω ότι έγιναν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα αυτά τα χρήματα από τα κράτη-μέλη και ήταν πολύ καλά όσον αφορά το, τη διασυνοριακή διάσταση Βερολίνο-Παλέρμο για παράδειγμα Μπρένερο, Λιόν-Τωρίνο Θέμα το οποίο συζητήθηκε ιδιαίτερα και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στον τύπο αυτή η σύνδεση Τωρίνο-Λιών. Πάντω χρηματοδοτήσαμε και, πολλά άλλα, και πολλά άλλα σχέδια. Και να σα πω επίση ότι χρηματοδοτήσαμε με ε, το πρόγραμμα ανάκτηση, το recovery plan, ε, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή και αποτέλεσε αντικείμενο χρηματοδότηση το περασμένο έτο, επενδύσαμε γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ για προγράμματα τα οποία μπορούσαν να εφαρμοστούν αμέσω ευθύ εκ αρχή ε, στα πλαίσια των δικτύων TEN, των διευρωπαϊκών δικτύων. Και αυτό λοιπόν είναι ένα άλλο σημαντικό μήνυμα για την σωστή χρήση των κοινοτικών κονδυλίων. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι οι επενδύσεις στα πλαίσια των διευρωπαϊκών δικτύων ε, είναι επενδύσεις που ακόμα και σε αυτή την ε, ε, περίοδο της κρίσης είναι πολύ χρήσιμα γιατί αφαιρούν τις υποδομές, γιατί θα δώσουν τη δυνατότητα ανάκαμψης, οικονομικής ανάκαμψης, θα δώσουν τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν μετρητά χρήματα για να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης ή τουλάχιστον να αναχαιτήσουν την ανεργία. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι καλέ επενδύσεις. Όσον αφορά τώρα ε, ε, του οργανισμού, ε, κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στι δύο μορφέ ε, γραφείων ή οργανισμών. Όσον αφορά του οργανισμού στα πλαίσια διαπρεπαϊκών δικτύων, όπω είπε και το ελεκτικό συνέδριο, νομίζω ότι λειτουργήσαν καλά και όσον αφορά την ικανότητα συνένωση μέσα στον ίδιο οργανισμό και σύγκληση συμφερόντων και αρμοδιοτήτων που ενδεχομένως ε, να είναι κάπως ε, ε, διχασμένα μεταξύ τους. Υπήρξε μεγαλύτερη προσέγγιση του πολίτη, μεγαλύτερη δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών και μάλιστα πρέπει να πω ότι απλοποιήθηκαν και πολλές γραφειοκρατικές πρακτικές. Και όπως ανέφερα, στις απαντήσεις που σας απέστειλα, εδώ είχαμε μία σειρά από θετικά στοιχεία, τα οποία προέκυψαν όσον αφορά ε, τις εργασίες ε, και τις, ΤΕΝ και τις ε, ε, ε, και του άλλου οργανισμού που διαχειρίζεται το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο. Επαναλαμβάνω, εξοικονόμηση χρημάτων. Γιατί υπήρξε εξοικονόμηση χρημάτων με το σύστημα αυτών των οργανισμών. Βελτίωση των υπηρεσιών, απλοποίηση των διαδικασιών, διαχείρισης, επαναλαμβάνω, μεγαλύτερη συνέργεια. Και είναι αλήθεια βεβαίως ότι στο κείμενο του, του, του ελεκτικού συνεδρίου προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση της σχέσης κόστους-οφέλους. Ναι. Και βεβαίως μπορεί να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση της εργασίας των οργανισμών αυτών. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο εμείς ε, το δεχόμαστε. Γιατί μπορεί να είναι καλή εργασία, αλλά πάντα μπορεί να βελτιωθεί ακόμα και ένα καλό αποτέλεσμα. Πάντω, όσον αφορά τι πτυχέ που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Επιτροπή σα, ε, τα γραφεία αυτά λειτουργήσαν καλά και προς το όφελος όλων ακόμα και από οικονομική άποψη. Θεωρώ λοιπόν την, ε, ε, ε απόλυτα θετικά τα αποτελέσματα και όσον αφορά την χρησιμοποίηση των δημοσίων χρημάτων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, αλλά σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο και την έκθεση του 2008 η κατανομή μεταξύ των γενικών διευθύνσεων ε, συμπεριλαμβανομένης της DigiTran, DG Γενικής Διεύθυνσης ε, ε, Περιφερειακής Πολιτικής δεν ήταν καλή και η το Ελεκτικό συνεδρίο λέγει ότι υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης μέσα στην Επιτροπή. Είστε αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να σχολιάσετε την παρατήρηση αυτή του Ελεκτικού συνεδρίου που αναφέρεται εις τις δαπάνες για έρευνα των μεταφορών, για έρευνα γενικώ, για θέματα συντονισμού, περιφερειακή πολιτική και ταμεία συνεχής όπου κατά 60% αφιερώνονται εις τις επενδύσεις για υποδομή μεταφορών. Και ε, υπάρχουν πολλοί λόγοι για ανικανοποίηση με την χρήση αυτών των χρημάτων. Επίσης ε, για τον, τη χρήση του, των πόρων του Ταμείου Συνοχής στις μεταφορές. Σαν αρμόδιος, μπορείτε να μας εξηγήσετε τις φράσεις αυτές τις οποίες έχει διατυπώσει το ελεγκτικό συνέδριο στην έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι τα κονδύλια για την έρευνα και η χρησιμοποίησή τους προέρχονται, ε, γίνονται ε, από διαφορετικές ε, υπηρεσίες επιτροπής με διαφορετικούς υπεύθυνου επιτροπούς. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ποτέ να μιλήσουμε για τέλειο συγχρονισμό των εργασιών, αλλά πρέπει να σας πω ότι από αντικειμενική άποψη και βεβαίω το ξαναλέω, κάθε καλό αποτέλεσμα μπορεί να βελτιωθεί και κάθε υπόδειξη του συνεδρίου για μένα είναι ευπρόσδεκτη. Γιατί αυτέ οι παρατηρήσει είναι χρήσιμε ε, και ε, προέρχονται από ένα θεσμό που αναπτύσσει θεμελιώδη ρόλο για τον έλεγχο. Και του ελέγχου, έλεγχο του ελέγχου που εμείς ε, με τη σειρά μας κάνουμε ε, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των δημοσίων χρημάτων. Πάντως γενικά πρέπει να σας πω ότι υπήρξε καλή συνεργασία ανάμεσα στους διάφορους τομείς ε, και τις υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι αρμόδιες για τα θέματα έρευνας. Εν μέρη απάντησα στην ερώτησή σας την ε, γραπτή ερώτηση υπαριθμών 8. Επαναλαμβάνω. Στην ε, απάντηση αυτή τη γραπτή, στην υπαριθμόν 8, επιβεβαιώνουμε ε, το γεγονός ότι είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε κάθε υπόδειξη του Ευρωπαϊκού του Ελεκτικού Συνεδρίου μέσα σε ένα κλίμα βέλτιστη συνεργασίας για την βέλτιστη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση των δημοσίων χρημάτων πιστεύουν θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή στρατηγική ε, ελέγχου, εξωτερικού ελέγχου, το είπα, και όσον αφορά τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορές. Στην γραπτή ερώτηση ε, μιλήσατε για ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με τα ε, μέσα πληροφορικής και κατά πόσον θα μπορούσε να είναι χρήσιμο ένα πιο αφιερωμένο μέσο πληροφορικής. Κοιτάξτε, ο συντονισμό και χάρη σε ε, όλες τις προσπαθειές μας αυτά τα χρόνια ε, είναι, ε, ενισχύθηκε ιδιαίτερα. Οι υπεύθυνε υπηρεσίε τη έρευνα προτιμούν μια λιγότερο τεχνική προσέγγιση που εκφράζεται συγκεκριμένα μέσα από διαρκείς συνεδριάσεις μεταξύ των διαφόρων υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για τους διάφορους τομείς έρευνας. Ορισμένα ζητήματα επί της ουσίας δεν είναι αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών. Αλλά και επαναλαμβάνω ότι η δέσμευσή μας είναι να φροντίσουμε έτσι ώστε να υπάρχει όλο και καλύτερη συνεργασία, όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, σε οργανωτικό επίπεδο, σε διοικητικό επίπεδο. Συνεργασία ανάμεσα σε εκπροσώπους των διαφόρων ε, γενικών διευθύνσεων που ασχολούνται με τα κονδύλια αυτά τα οποία ε, προορίζονται για την έρευνα. Όταν θα ο επίτροπο για θέματα ε, βιομηχανίας, και εκεί θα διαχειριστούμε κονδύλια που έχουν στόχο την έρευνα και εκεί θα συνεχίσουμε τι προσπαθίε μα για να αποδείξουμε συνολικά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εργάζεται με τον βέλτιστο τρόπο, όχι μόνο σε τεχνικό και γραφειοκρατικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, για να ελέγχουμε έτσι ώστε και ε, απέφχομαι ε, κάτι τέτοιο ε, στην περίπτωση απάτη, αν θέλετε. Θέλουμε να υπάρχουν όσο και, με, και λιγότερε απάτε, αλλά και όσον αφορά κακή χρησιμοποίηση των χρημάτων. Και να έχουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερο κατόφλι σφαλμάτων όταν μιλάμε για χρησιμοποίηση και αξιοποίηση δημοσίων χρημάτων. Σα ευχαριστώ, κύριε Λιμπεράς. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Ο χρόνος είναι περιορισμένος και θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα στους συναδέλφους. Έχουμε 30 λεπτά. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι. Κύριε Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, Καλό είναι που θα παραμείνετε στο χειρισμό της, ε, ε, του φακέλου Γαλιλαίου διότι φεύγετε από τις μεταφορές και τον παίρνετε μαζί σας οπότε θα έχουμε επαφή επ' αυτού. Θα ήθελα να αναφερθώ ή στη συσσόρευση των ε, μέσων διότι το Γαλιλαίο χρηματοδοτήθηκε και εις βάρος των ε, του Γεωργικού Ταμείου ε, αλλά υπέρ της βιομηχανίας. Τότε όμως είχαμε αμφιβολίες εάν θα έφταναν τα χρήματα και τώρα είπατε ότι θα χρειαστείτε ακόμη περισσότερα χρήματα. Είναι κάτι το οποίο ήξερε ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε ότι χρειαζόταν περισσότερο χρήματα. Όντως ισχύει αυτό ή τι ήταν η κατάσταση σχετικά με ε, αυξημένη ανάγκη πόρων. Επίσης όσον αφορά τους φακέλους. Το Γαλιλαίο είναι ένα μπαλάκι που άγεται και έρχεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, το να παραμείνει εις τις μεταφορές έχει ε, νόημα, αλλά αυτή τη στιγμή έχει μεταφερθεί στη βιομηχανία όπου έχει περιορισμένες δυνατότητες. Ε, δηλαδή ε, τι άνθρωποι θα χρειαστούν από πλευράς οικονομικού ελέγχου για να διασφαλιστεί η σωστή πορεία του Γαλιλαίου στο μέλλον. Επίσης αναφερθήκατε στην συνεργασία με την ΕΖΑ. Έχετε την πρόσβαση στα στοιχεία όταν την επιθυμείτε ή βασίζεστε απλώς σε παραστατικά της ΕΖΑ. Πώς λειτουργεί το σχετικό σύστημα ελέγχου. Και τέλος για τη Βουλγαρία όπου υπάρχει ένα γραφείο ε, για το δικό σύστημα όπου είχαν ε, διατεθεί πόροι το 2009 για το, ε, την τον Ιουλιανό αυτοκινητόδρομο όπως λέγεται Ιουλιανό το Way θα ήθελα να ξέρω τι έγινε με τα προβλήματα που αντιμετώπισε ε, και αν είστε ικανοποιημένος με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων που έχετε στον τομέα σας διότι ε, έχουμε 3-4 δισεκατομμύρια για τον Γαλιλαίο και 900 ε, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κέρδος αν όντως είναι τα πράγματα σας συγχαίρω. Πρόεδρε, για μια μισή ώρα θα μπορούσα να μιλάω για αυτά τα θέματα, έτσι. Α, πέντε λεπτά. Όχι, εντάξει, αστειευόμουν. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομο. Όσον αφορά το Γαλιλαίο, στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα έδωσε νομική βάση για μια πολιτική στο τομέα του διαστήματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πρόεδρο Μπαρόζο θεώρησε σκόπιμο ε, να ε, ανατεθούν όλα αυτά σε ένα και μόνο επίτροπο. Γιατί ξέρετε ότι εκτό του Γαλιλαίου και του Έγνωσου. Έχουμε το, το πρόγραμμα GMS που αφορά κυρίως σε την διαστημική πολιτική που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Έχουμε το έγνος βεβαίως και βεβαίως, όπως προβλέπεται και από τη συνθήκη, έχουμε, μια, έχουμε τη δυνατότητα για ένα διαστημικό πρόγραμμα έρευνα και ανακάλυψη, αν θέλετε, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η απόφαση του Πρόεδρου Μπαρόζο ε, να τα αναθέσει όλα αυτά σε έναν και μόνο επίτροπο και δεδομένη ε, τη ε, βιομηχανική σημασία. Και επειδή εδώ υπάρχει αλληλοσύνδεση των διαφόρων συστημάτων του GMS και το Γαλιλαίο, κυρίως ως προς τις ε, κοινωνικές πτυχές και επιπτώσεις. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η σύζυξη ήταν κρίσιμη. Τώρα, να σα πω για αυτά που ξέρω από τι 9 Μαου του 1998, από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Στο, ε, προηγουμένως ως μέλος του Κοινοβουλίου ήξερα αυτά που ξέρετε κι εσείς. Αν υπήρξαν ορισμένα πράγματα απόρριτα δεν τα ξέρω εγώ. Πάντως μπορώ να σας πω όσον αφορά τα κονδύλια. Ότι τα κονδύλια ε, για το σκοπό αυτό είναι 3,9 δις ευρώ. 3,6, Ζητώ συγγνώμη λέει ο Επίτροπο. 3,6 δι. Θα υπάρξει αύξηση. Εγώ δεν είπα ότι αναπόφευκτα θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα και ότι θα υπάρξει αίτημα για περαιτέρω κονδύλιο. Το μόνο που είπα ήταν ότι όσον αφορά αυτά που έχουμε προγραμματίσει για ε, τις απαντήσεις, κτλ. Ε, ε, βρισκόμαστε με του προπολογισμού. Είπα ότι δεν αποκλείω όταν μετά το 2014 θέλουμε να φτάσουμε και κοιτάξτε Βεβαίω, η πρόβλεψη θα γίνει εκ των προτέρων. Αν δούμε ότι απαιτούνται περαιτέρω κονδύλια, δεν ξέρω. Ούτε καν μπορώ να σα πω για ποιο νούμερο μιλάμε. Θα ήταν ε, ε, ε, επιπόλαιο να κάνω κάτι τέτοιο. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με πτυχέ που αφορούν την έρευνα, τεχνικά ζητήματα κτλ. Πάντω, σα είπα, ε, και το είπα και στου συναδέλφου όταν έκανα την ακρόαση ως υποψήφιο επίτροπος ε, βιομηχανία, ε, αναλαμβάνω επίσημα τη δέσμευση και με τι δική τη επιτροπή, Πρόεδρε, να έρθω και να ενημερώσω το Κοινοβούλιο. Μόλις έχω κάτι χειροπιαστό στα χέρια μου. Μόλι έχω κάποια αξιόπιστα στοιχεία για το ότι θα απαιτηθούν για παράδειγμα, νέα κονδύλια, σα λέω δεν το αποκλείω. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σα πω ότι ναι, θα χρειαστούμε χίποσο. Μπορούμε να σας πω με βεβαιότητα ότι αυτό το οποίο ήδη έχουμε προβλέψει ε, μέχρι το 2014 ε, φτάνει μέχρι το 2004. Όσον αφορά τη Βουλγαρία τώρα, δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Τα προγράμματα και τα σχέδια τα οποία αναφέρθηκαν από την κυρία Γκρέσε αφορούν ε, περιφερειακά κονδύλια. Εμείς ε, δεν έχουμε χρηματοδοτήσει κάτι τέτοιο στη Βουλγαρία ε, στα πλαίσια του NT. Δεν, δεν είμαι σε, φάση, λοιπόν, σε θέση συγγνώμη, να σα δώσω κάποια απάντηση. Πρέπει να ρωτήσετε τον αρμόδιο επίτροπο. Όσον αφορά τη σημασία, ε, τι να σας πω, θα μπορούσα να παραταθώ και να μακρηγορήσω για πολύ. Όσον αφορά ε, την ε, σημασία του Γαλιλαίου, μπορώ να σας πω πολλά, αλλά ίσως θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ερωτήσεις. Η κυρία Γιάννα Σέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε, για το Γαλιλαίο ε, που μας απασχολεί σήμερα και γιατί πρόκειται για ένα θεμελιώδες ε, σύστημα το οποίο θα μας γλιτώσει από πολλά δεινά. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα που θα πάτε λοιπόν στη βιομηχανία μου έρχονται στο μυαλό δύο ερωτήσεις. Κύριε Ταγιάννη, που βεβαίως να σας πω ότι έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στι ικανότητε σα πω ότι εσεί θα έχετε αρκετά κονδύλια ε, στη βιομηχανία, γιατί ε, βεβαίω τα δίκτυα θα απαλλαγούν από το Γαλιλαίο. Μεγάλο το βάρο το οικονομικό. Αλλά θα βρείτε χρήματα στη βιομηχανία για το Γαλιλαίο. Ε, με βάση τη διαστημική πολιτική που είπατε κι εσεί. Τι θα γίνει, ε, η βιομηχανία θα την αναλάβει τη χρηματοδότηση, γιατί εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Και δεύτερον, όσον αφορά με αυτά τα οποία διαβάσαμε στον τύπο. Να σα ρωτήσω το εξή, γιατί εδώ υπάρχει μια διαδικαστική, ένα διαδικαστικό ζήτημα το, στο οποίο προσκρούμε διαρκώ. Δηλαδή, μέχρι να ολοκληρώσει, ε, ε, από τη μια έχουμε να, να περιμένουμε να ολοκληρώσει την εξέτασή του ε, το, ε, το δικαστήριο και από την άλλη να δούμε τι θα γίνει. Το ελεκτικό συνέδριο, δηλαδή τι θέλω να πω. Ε, όταν κάνει την πρώτη ε, ε, την πρώτη παρέμβασή του το, το συνέδριο, ε, όταν έκανε την πρώτη παρέμβαση το συνέδριο, είπε το Γαλιλαίο ήταν σε κρίση, αν μπορώ να το πω έτσι. Τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο τη υλοποίηση. Θέλω λοιπόν να σα ρωτήσω για άλλη μια φορά επί τη διαδικασία. Όσον αφορά τη συνεργασία ε, του ελεκτικού συνεδρίου ε, με την Επιτροπή σε σχέση με τις προθεσμίες. Τώρα, κοιτάξτε, ε, εγώ είμαι η συγγήτρια για το ΦΕΔ σε σχέση με τον κύριο Λιντεράσκι, που είναι ο βασικός εισηγητής για την απαλλαγή. Σας ρωτώ λοιπόν, εσείς πράγματι, και σας χαίρω γι' αυτό, καταβάλλετε σημαντική προσπάθεια για τα δίκτυα στα πλαίσια ε, της ε, ε, Μεσογείου και της ε, ε, με την περιοχή αυτή. Στείλετε κάποιους υπαλλήλους από την Γενική Διεύθυνση Τρέν και τα λοιπά. Ναι, θέλετε να δώσετε πολιτική όθηση. Ρωτώ όμως, πώς συνδέονται αυτά ε, τα θέματα που έχουν ε, ε, να κάνουν με τα κονδύλια της Γενικής Διεύθυνσης Τρέν που αφορούν ακριβώς την πολιτική γυπνίασης με τα υπόλοιπα στοιχεία. Με τα, με υπόλοιπα προγράμματα, με έντα κτλ. Υπάρχει καλός συντονισμός ή πρέπει να γίνουν κι άλλα και πρέπει, εμείς να, πρέπει να δώσουμε περαιτέρω όφηση από άποψη δική μας επιτροπή. Και τέλος, όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τώρα εμεί προσπαθούμε να υποχρεώσουμε κατά κάποιο τρόπο τα κράτη-μέλη να αναλάβουν την ευθύνη ενώπιον του Κοινοβουλίου, να είναι υπόλογα ενώπιον του Κοινοβουλίου και ενώπιον τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση, συγχρηματοδότηση. Όσο, με βάση τη δική σα εμπειρία στη Γενική Διεύθυνση Τρέν, πώ μπορούμε να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να, να συγχρηματοδοτούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Θα υπάρξει κάποιο μέσο, κάποια συγκεκριμένη διαδικασία για να αναγκάσουμε κατά κάποιο τρόπο τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τι ευθύνε του. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένε συμφωνίε, αλλά ποτέ δεν υπάρχει ε, απαραίτητο απαραίτητο βαθμό χρηματοδότηση. Κυρία Γιάννα θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Η συνεργασία μας με το Κοινοβούλιο και με το Ελληνικό Συνέδριο και το Συμβούλιο απαιτείται και είναι χρήσιμη για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Καταφέραμε και επειδή το ζήτησε το ελεκτικό συνέδριο αλλά και με συνεχή σχέση ελέγχου που ασκεί, πολιτικό έλεγχο που ασκεί στο έργο της Κομισιόν το Κοινοβούλιο και γι' αυτό το πρόγραμμα είναι κοινοτικό. Χρηματοδοτούν και τα κράτη-μέλη αλλά στην Κομισιόν με το, στον κοινοτικό προπολογισμό από εκεί ξεκινάνε όλα αυτά. Αυτή η στενή συνεργασία όλων μας λοιπόν μας επέτρεψε να διορθώσουμε λάθη και να κάνουμε πιο αποτελεσματική τη δουλειά μας και τη συνεργασία μας ειδικά με το Ελεκτικό Συνέδριο άριστη, αγαστή η συνεργασία. Και όταν υπήρξαν αιτήματα για διευκρινήσεις ή υποδείξεις και προτάσεις εμείς πάντα δεχτήκαμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό να τα ικανοποιήσουμε όλες τις υποδείξεις και όσον αφορά το λογιστικό σκέλος και όσον αφορά τους ελέγχους για το δημόσιο χρήμα. Γιατί πιστεύω ότι όλα αυτά είναι χρήσιμα. Όπως επίσης και ο πολιτικός έλεγχος. Τώρα η σχέση του Γαλιλαίου με τα δίκτυα TEN. Το Γαλιλαίο είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα που θα μας απλουστεύσει τη ζωή. Δέστε πώς άλλαξε ε, με τη χρήση του GPS τα συστήματα γεωπλοήγησης. Έχουμε ένα αυτοκίνητο, έχουμε μπροστά ένα, μια μικρή οθόνη που μα επιτρέπει να πάμε όπου θέλουμε. Σκεφτείτε πόσε άλλε χρήσει μπορεί να έχει ότι θα μπορούμε να παρεμβαίνουμε με σινιάλα που θα μα έρχονται από του δορυφόρου και το σύστημα Γαλιλαίου για να σώσουμε ανθρωπινε ζωέ ή για να παρέμβουμε σε διάφορε άλλε τραγωδίε. Σκεφτείτε ένα δορυφορικό ευρωπαϊκό σύστημα, όλες οι, η άμεση βοήθεια που να συντονίζεται για την ΑΕΤ Φερρυπίνο, ότι πάει το υλικό, να χρησιμοποιούν υλικό που προερχόταν από το Ευρωπαϊκό Δορυφορικό Σύστημα. Και αυτό έγινε, είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που μας δείχνει πως ορισμένα συστήματα μπορούν να είναι χρήσιμα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό για την Αφρική, να χρησιμοποιήσουμε τα δορυφορικά ευρωπαϊκά συστήματα. Γιατί το Γαλιλαίο είναι τμήμα είναι ο πιο σημαντικός αδελφός, πιο μεγάλος αδελφός ας πούμε ενός συστήματος που έχει το έγνος, το GMS και όλη η δουλειά που έγινε στο παρελθόν μέχρι σήμερα σε συντονισμό και με μη ευρωπαϊκά προγράμματα του GPS Φερρυπίν. Τα ευρωπαϊκά συστήματα βοηθάνε παραδείγματος να προσαρμοστούν σινιάλα που θα, χάρη στο έγνος θα κάνουν πιο εύχριστα τα μικρά αεροδρόμια στην Ευρώπη. Σήμερα πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται μόνο την ημέρα. Χάρη στα σινιάλα GPS από το έγνος και μετά από το γαγγελέο θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε 24 ώρες το 24ωρο μικρά αεροδρόμια. Για τους χρήστες. Μετά την τελευταία έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου χρησιμοποίησαμε ορισμένα εργαλεία, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, ε, προγράμματα που έχουν προτεραιότητα, νέο οικονομικό ε, κανονισμό, η σχετική υπηρεσία που υπάρχει. Η κυρία Γιάλα Σέντερ ξέρει γιατί έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν να συζητήσουμε για το θέμα των συντονιστών που είναι ουσιαστικά η φωνή της Κομισιόν προκειμένου να πιστούν τα κρατημέλη να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά κολλήματα, ιδιαίτερα στα σύνορα και οι χώρες να τηρούν τις υποχρεώσεις που έχουν πάρει και αυτοί και εμείς και μεταξύ μας. Επενδύουμε κοινοτικά χρήματα και κονδύλια. Αν το κράτος μέλος δεν επενδύσει και αυτό το μερίδιό του, ε, καταπίπτει όλο το σύστημα, καταπίπτει η επένδυση. Έχουμε λοιπόν την υποχρέωση εμείς να είμαστε αυτός που θα κατευθύνει την επένδυση. Η δική μας επένδυση, ελπίζω, να ε, συσπυρώσει κονδύλια και των κρατών μελών και ιδιωτικά. Και ιδιωτικά, το τονίζω αυτό. Αυτά έχουν γίνει και ορισμένες διορθώσεις επίσης έχουν γίνει όπως τα ζήτησε το συνέδριο για την 2007 2013 η δυνατότητα να παίρνονται αποφάσεις για χρηματοδότηση πολυετή. Οπότε ο έλεγχος μπορεί να γίνεται συνεχής και ad hoc και οι αποφάσεις της Κομισιόν μετά την ψήφο της Οικονομικής Επιτροπής και με βάση τα τη νομοθεσία όπως έχει οριστεί από τη μεριά του Ευρωκοινοβουλίου μας επιτρέπουν στενή συνεργασία με την εκτελεστική υπηρεσία και τους δικαιούχους, δηλαδή τα κράτη-μέλη. Άρα αυτό που λέει η, η κυρία Αγιάλα είναι, ένα, είναι και δικός μας προβληματισμός και θα φροντίσω τα κράτη-μέλη να τηρούν τις υποχρεώσεις τους ως Επίτροπος Μεταφορών. Τώρα, για τη χρηματοδότηση για το Γαλιλαίο μέχρι το 2013. Μετά θα δούμε. Αναφερθήκατε στην αλλαγή κατεύθυνσης. Η χρηματοδότηση του Γαλιλαίου είναι ε, διαφορετικό από τη χρηματοδότηση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. με τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Μην ανησυχείτε ιδιαίτερα γιατί ότι υπάρχει το πέρασμα από τις μεταφορές στη βιομηχανία. Εγώ πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να έχουμε μια ενιαία πολιτική για το διάστημα. Δεν είναι μόνο ο Γαλιλαίο, είναι όλη η πολιτική του διαστήματος την οποία συζητάμε εδώ και στην οποία ευτυχώς η συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε νομική βάση. Ο κύριος Γκέιερ. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι ε, ε, πολλά δεν είπε ο πρόεδρος αλλά ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αλλά δεν έχουν πολύ χρόνο ε, αναφερθήκατε σε αύξηση του κόστους για τον Καλλιλέο όλοι γνωρίζουμε ότι τον Καλλιλέο θα είναι μία πρόοδος διότι δεν θα έχει δεχθεί διαφορετικά το Κοινοβούλιο μέχρι τώρα τις αυξήσεις των δαπανών αλλά το ερώτημά μου είναι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω στο Γαλιλαίο και αν όχι πώς θα αντιμετωπίσετε την βιομηχανία που ζητά αύξηση των πιστώσεων για τον Γαλιλαίο δηλαδή πώς, πώς θα εμποδίσετε να υπάρχουν άλλες απαιτήσει από τη βιομηχανία για να μπορέσει αυτό το πρόγραμμα να εξυπηρετήσει την ε, διαστημική έρευνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κατάλαβα πολύ καλά. Την απάντηση όμως θα τη βρείτε στην απόφασή μας πριν από μερικές εβδομάδες όπου αποφασίσαμε να δώσουμε θετική απάντηση στις επιχειρήσεις που, των οποίων οι προτάσεις ήταν κάτω από την οροφή. Δηλαδή, φροντίσαμε με τη Γενική Διεύθυνση και με την υπηρεσία, όπως είπα και πριν, σχέση, ποιότητα, τιμή. Τα λεφτά δηλαδή να πιάνουν τόπο. Και επειδή υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, άλλες είναι για τους δορυφόρους. Μερικοί δορυφόροι γίνονται από μία εταιρεία που δεν ε, προκρίθηκε στο διαγωνισμό πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτό είναι απόδειξη ότι η Κομισιόν δεν θα υποκύψει σε αιτήματα της βιομηχανίας λέγοντας να, μπορούν, να μπορεί να έρθει και να μας πει αν θέλετε να κάνετε προγράμματα πρέπει να μας δώσετε λεφτά. Φυσικά προβλέφτηκαν ορισμένε αυξήσει. Εξάλλου με τα φιλόδοξα τέτοια προγράμματα αυτό συνήθως γίνεται. Πάντως εμείς δεν πρόκειται να εκβιαστούμε από κανέναν. Δέστε τον τελευταίο διαγωνισμό και πώς δόθηκαν τα έργα. Τηρήθηκε 100% με αυστηρότητα, με πολλές ώρες συζήτησης για την κάθε παρτίδα, για τον κάθε αντικείμενο του διαγωνισμού προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να είναι σεβασμός στη χρήση των χρημάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Η πολιτική μου βούληση είναι να μην ενδώσω σε καμία περίπτωση σε εκβιασμούς ή σε καταστάσεις μονοπωλίου. Ο ανταγωνισμός να λειτουργεί και βοηθάει την καλή ποιότητα του προϊόντος, χωρίς βάρος όμως κανενός ή προτιμώντας κάποιον τρίτον. Το πρόγραμμα ήδη είναι προχωρημένο. Σας είπα ότι το 2014 είναι το έτος κλειδί που θα αρχίσει να λειτουργεί ο Γαλιλαίο. Αν θέλουμε, πέραν αυτού του έτους, να συμπληρώσουμε το αρχικό πρόγραμμα, δηλαδή να αναπτυχθούν όλοι οι δορυφόρε για να λειτουργεί όπως προβλεπόταν στο αρχικό σχέδιο στην περίπτωση αυτή είναι πιθανό να χρειαστεί να ξανάρθουμε στο Κοινοβούλιο και να σας πούμε ξεκινάει το πρόγραμμα αλλά αν θέλουμε από κοινού τα τρία θεσμικά όργανα να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα όπως είχε προβλεφθεί στην αρχή χρειαζόμαστε αυτά τα ποσά. Επαναλαμβάνω, το είπα στην Ακρόση και το ξαναλέω και ευχαρίστω όποτε με ξανακαλέσετε να ξαναρθώ να σα απαντήσω. Εγώ θα πάρω πρωτοβουλία και θα σας πω. Σήμερα, σήμερα σας λέω την πολιτική αξιολόγηση που έχουμε κάνει. Δεν μπορώ να σας δώσω λογιστική, οικονομική εικόνα. Δεν μπορώ σήμερα. Πολιτική αξιολόγηση, ναι. Μετά από κοινού αργότερα θα ορίσουμε τι οικονομική και λογιστική απάντηση θέλουμε να δώσουμε στο πρόβλημα. Πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, έχω κι εγώ μια ερώτηση. Στο σημείο 4 της απάντησής σας, Λιόν Τωρίνο, μπορείτε να μας πείτε κάτι για το κόστος πέραν της περίοδου γιατί είπατε ότι οι δικαιούχοι δεν είχαν δικαίωμα αλλά ήταν καλόπιστοι λοιπά Μπορείτε να μας το ξεκαθαρίσετε λίγο παραπάνω αυτό το σημείο 4. Αφορά το 2004-2005 κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριο Σταγιάννη. Ήταν ένα τυπικό λάθος. Δηλαδή το συγκεκριμένο κράτος μέλος υπέβαλε ένα αίτημα. Μια γραφειοκρατική οργάνωση του παρελθόντος μέχρι τότε δεν, πήρε θετική απάντηση να παραταθεί η προθεσμία. Τα κονδύλια δόθηκαν με βάση το αίτημα του κράτους μέλους. Δεν υπήρχε κακοπιστία. Τα ποσά ήταν δεδομένα. Κατά τη γνώμη μας η απάντηση έπρεπε να είναι ναι εκ μέρους της Επιτροπής. Γραφειοκρατικό λάθος ήταν. Ας πούμε η επιστολή καθυστέρησε κάπου που δεν έπρεπε να καθυστερήσει να μπλοκαριστεί. Δεν υπήρχε ούτε δόλος, ούτε ιστεροβουλία. Ένα γραφειοκρατικό σφάλμα. Επαναλαμβάνω, γραφειοκρατικό σφάλμα αλλά όχι δόλος ούτε εκ μέρους της κυβέρνησης ούτε εκ μέρους της Επιτροπής. Έλειπε η απαντητική επιστολή που, λέει, που έλεγε ναι σας δίνουμε την παράταση γιατί έχετε το δικαίωμα στην παράταση. Περί αυτού πρόκειται. Δόλος μηδέν. Ούτε απάτη ούτε κακή προαίρεση, ούτε η προσπάθεια κατάχρησης των κοινοτικών κονδυλίων εκ μέρους της χώρας. Γκρέσλερ. Ήθελα να σας υπενθυμίσω το θέμα που έχει μείνει ανοιχτό. Δηλαδή πώς μπορούμε να ελέγξουμε την ΕΖΑ, την Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διαστήματος. Τι στοιχεία υπάρχουν για αυτό το στόχο. πώς ελέγχουμε τις προσφορές που γίνονται σε σχέση με τις ε, ε, προκηρύξεις διαγωνισμών. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε αναθέσει στον οργανισμό διαστήματος να ε, ασχοληθεί με την εργασία αυτή. Η τελική απόφαση βεβαίως ανήκει στην Επιτροπή. Όσον αφορά αυτές τις τελευταίες τρεις παρτίδες, έφτασε σε μένα ε, η εργασία της, ε, του οργανισμού, εργαστήκαμε πάνω στο θέμα αυτό, είδαμε τη σχέση κόστος-οφέλους, ε, ανώτατα όρια της Επιτροπής, ε, ε ανώτατα όρια σε σχέση με ορισμένε προτάσεις που έγιναν από τους διαγωνιζόμενους. Ελέγξαμε, το ξαναλέω, τη σχέση ποιότητας τιμής και, επειδή, και βεβαίως στα πλαίσια ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μονοπόλια, προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πολιτών. Τώρα, ε, όσον αφορά ε, τη σύμβαση θεσπίζεται από, την, ε, από τον οργανισμό και όταν περνάμε από τη φάση της έρευνας στην επιχειρησιακή φάση ε, το, το Γαλιλαίο όπως και με το έγκνος θα περάσει στον ε, απευθείας έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως και το τμήμα το οποίο αφορά την κινητοποίηση αυτή θα έρθει στην Επιτροπή. ε, τον προπολογισμό 2009 θα ε, συμπεριληφθεί και το έγνος, γιατί το έγνος ε, από φέτος ε, έφτασε στην άμεση, πέρασε στην άμεση διαχείριση επιτροπής. Όταν θα έχουμε και την, τελειώσει και η φάση της έρευνας στο Γαλιλαίο, το ίδιο θα γίνει και στην περίπτωση αυτή, θα ενταχθεί στον προπολογισμό της Επιτροπής. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. υπήρξε αυτή η συμφωνία για την ανάθεση στην, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματο. Απαντώ και στην προηγούμενη ερώτηση. Βεβαίω, ε, ό,τι ζητάμε μας, δίνεται, όλα τα στοιχεία μας τα δίνει, η υπηρεσία κτλ. Και όταν τους προσκαλούμε έρχονται και συνεδριάσει τη οργανική ομάδα, Επιτροπή, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο που ε, συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ε, Βεβαίω ε, μπορούμε να βάλουμε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια στα πλαίσια τη διοργανική ομάδα να, δώσουμε, να δώσουμε στην ομάδα αυτή ε, ε, περισσότερο βάρο και περισσότερε δυνατότητε ε, ακριβώ για να αντιμετωπίζονται οι λεπτομέρειε των διαφόρων ζητημάτων επειδή στην προηγούμενη μου ζωή ήμουν δημοσιογράφος, καταλαβαίνετε ότι έχω την, ε, ε, αυτή την ε, περιέργεια, σκαλίζω τα πράγματα, προσπαθώ να δω τι βρίσκεται από πίσω. Ελπίζω λοιπόν αυτή η δραστηριότητά μου, η ερευνητική μου δραστηριότητα εντό εισαγωγικών, να είναι χρήσιμη. Πάντω έχω την εντύπωση ότι ο οργανισμό πάντα ε, ανταποκρίθηκε με σαφήνεια στα δικά μα τα αιτήματα. Και το ξαναλέω, είμαι έτοιμο βεβαίω να δεχτώ και τι τυχόν υποδείξει ε, έχετε όλη την ε, ευχαίρεια να υποβάλλετε ερωτήσει, αν έχετε αμφιβολίε. ακόμα και ανεπίσημα πέραν ε, των ερωτήσεων που τίθενται στη διοργανική ομάδα και ε, στην ακρόαση και σε ανεπίσημη βάση. Είμαι έτοιμο να, έρθω, σε επαφή μαζί σα, να συναντήσω, αν θέλετε, συγκεκριμένε διασαφηνήσει. Ε, Βεβαίω μπορείτε και μέσω εμού να τα υποβάλλετε τα ερωτήματά σα στον οργανισμό διαστήματο, ε, στην υπηρεσία διαστήματο. Μέγιστη διάθεση και μέγιστη διαφάνεια. Να δώσουμε σύντομα το λόγο στην κυρία Γκλέφτελε. Ίσως δεν έχετε καταλάβει το νόημά μου και θα το εξηγήσω. Έχουμε πολλών ειδών χρηματοδοτήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ε, πώς ε, σκέφτεται κανείς να χρησιμοποιήσει ένα πρότυπο χρηματοδότησης για την ΕΖΑ. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ε, πώς είστε βέβαιος ότι είναι σωστό το σύστημα χρηματοδοτήσεως. Έχουμε ενωμένα Έθνη παραδείγματος χάρη εκεί μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Θα θέλω όμως να ξέρω πώς εσείς είστε βέβαιος από τους εξωτερικούς ελεγκτές ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος είναι, πηγαίνει καλά. Πώς γίνεται η, σωστή, η χρηστή διαχείριση δηλαδή. Ευχαριστώ. Επειδή ε, ε, εκτός, ο πρόεδρο συνεχίζει εκτό μικροφώνου. Μάλιστα. Επειδή είναι τελευταία ερώτηση προ τον Επίτροπο και επειδή εμεί και στι προηγούμενε συνδράσει είχαμε αναφερθεί στον Γαλιλαίο, όπω καταλαβαίνετε κι εσεί ε, και προφανώ το ενδιαφέρον μα είναι τεράστιο και επικεντρώνεται στη διαφάνεια, όπω είπατε κι εσεί, στο πώ δαπανώνται τα χρήματα προ το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών και φορολογουμένων. Έχουμε λοιπόν την ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε ε, που αφορά και τις διαδικασίες ανάθεσης, διαδικασίες των ε, δημοπρατήσεων. Τι δεσμεύσεις αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ενώπιον της δικής μας Επιτροπής. Είναι η τελευταία ερώτηση που σας γίνεται. Επίτροπε, έχετε το λόγο. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή η συνεργασία είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Τι δεσμεύσεις αναλαμβάνω ενώπιον του Κοινοβουλίου, τι να σας πω. Ε, ήμουν μέλος για 15 χρόνια. Οι δεσμεύσει αυτές ε, αφορούν όχι μόνο το επίσημο επίπεδο, σας το είπα, αλλά σας το λέω και άλλη μια φορά. Ό,τι έγγραφα χρειάζεστε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να σας το δώσουμε. Ε, σε οποιοδήποτε μέλος ε, της Επιτροπής σας. Όπως είπα και στην απάντηση ε, υπαριθμών 2, στη γραπτή μου απάντηση. Παραθέτω όλες τις συμφωνίες που συνάψαμε με την ε, υπηρεσία, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Εκεί δώσαμε, κάναμε τη συγκεκριμένη ανάθεση καθηκόντων για την επεξεργασία ε, της, ε, της, του, σταδίου της έρευνας και, για την αξιολόγηση των προσφορών. Δηλαδή, το ξαναείπα, η τελική απόφαση έγκυται σε εμά. Τη σύμβαση όμω την υπογράφει η υπηρεσία. Νομίζω ότι αυτό είναι θετικό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουμε και το εξωτερικό στοιχείο το οποίο επισέρχεται. Ακούσαμε τις επικρίσεις ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου και αλλάξαμε τον τρόπο συνεργασίας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΕΖΕ λοιπόν ε, είναι ένας οργανισμός της Επιτροπής στην οποία εμείς δίνουμε input. Το ξαναλέω. Μετά από τη φάση της έρευνας το Γαλιλαίο θα ξαναγυρίσει στον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον άμεσο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ό,τι έγραφο λοιπόν θέλετε κυρία Γκρέσε. κυρία Γκρέσλε, πολύ ευχαρίστω θα σας το δώσω. Θα φροντίσω να το πάρετε. Αν χρειάζεται θα ζητήσω από την υπηρεσία διαστήματος αυτά τα στοιχεία που θέλετε να δείτε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι εκ μέρους της υπηρεσίας διαστήματος υπήρξε μέγιστο επίπεδο συνεργασία και έναντι του Κοινοβουλίου. Γιατί οι εκπρόσωποι τη υπηρεσία ε, νομίζω ότι πάντα έρχονταν, όχι μόνο επίσημα, αλλά και ανεπίσημα ε, και σε επίπεδο ε, διοργανική και ομάδα εργασία συμμετείχαν ιδιαίτερα επικοδομητικά, έδιναν στοιχεία και πάντα μιλούσαν για το πού βρισκόμαστε. Επειδή ήρθαν πριν από την ανάθεση των τελευταίων τριών παρτίδων, νομίζω ότι έγιναν δύο-τρει συνεδριάσει όπου δόθησαν στους προσώπους του Κοινοβουλίου όλες οι διασαφηνήσεις και όλες οι πληροφορίες. Καθώς και τα στοιχεία τα οποία ζήτησαν τα μέλη του Κοινοβουλίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και αν θεωρείτε και εσείς σωστό, Πρόεδρε, κοιτάξτε, έχουμε τη διοργανική ομάδα που αποφασίζει ποιος ε, ε, για την εκπροσώπηση. Πάντω, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, πρόεδρε. Να έρχομαι στα 7 χρονικά διαστήματα, όποτε το θέλετε. Όπου θέλετε σκόπιμο, να έρχομαι να σα ε, ε, λέω τι γίνεται για το Γαλιλαίο. Στα πλαίσια τη μέγιστη διαφάνεια, το λέω, το επαναλαμβάνω, κύριε πρόεδρε. Και αν θέλετε σκόπιμο, ε, και έχετε και την καλοσύνη να μου, να μου γνωστοποιείτε εκ των προτέρων τι ε, έγγραφα θέλετε να δείτε, εγώ θα φροντίσω είτε δημόσιο είτε κατηδίαν ό,τι θέλετε. Θα, θα να σα δώσω το έγγραφο που θέλετε. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Επίτροπο Ταγιάννη. Και τώρα νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε ε, με, την, με τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσια διάταξης. Έχουμε πολλά θέματα ακόμα μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στη χορήγηση απαλλαγή του 2008 όσον αφορά τους οργανισμούς. Ιδιαίτερα για την Ευρωπαϊκή Αστυνομία, Αστυνομική Ακαδημία, ΣΕΠΟΛ και για το Frontex, Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση Επιχειρησιακή Συνεργασία στα εξωτερικά Συνέδρια των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δώσω το λόγο στο μέλο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, Νατζέντα Σαντολόβα. Okay, thank you very much. It was nice. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού, εν ονόματι του Ελεκτικού Συνεδρίου, έχω τη χαρά να παρουσιάσω ε, την ε, θέση των Ευρωπαϊκών Οργανισμών για τους ε, λογαριασμούς του 2008, όπου το συνέδριο έχει ελέγξει 29 οργανισμούς, εκ των οποίων 25 ρυθμιστικοί και 4 εκτερεστική. Ο προπολογισμό είχε σύνολο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για το ε, έτος 2008. Δύο γραφεία, ε, το γραφείο στην Ονζέ και το γραφείο εναρμονίσεως εσωτερικής αγοράς στην Αλικάντε έχουν ε, χωριστεί απαλλαγή από τις δημοσιονομικές τους αρχές. Τώρα θα αναφερθώ εις δύο ο οργανισμούς των οποίων εκπρόσωποι έχουν κληθεί εδώ. Το 2007 το Συμβούλιο θεώρησε ότι δεν υπήρχε ένα σωστό σύστημα δεσμεύσεων. Κατά τον έλεγχο του 2008 διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν δυσκολίες μεταφοράς στο νέο λογιστικό σύστημα BAC στην ε, εφαρμογή ε, του συστήματος δεσμεύσεων ε, που προκαλούσε υπερβολικές καθυστερήσεις και στην έγκαιρη πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού που δεν προχωρούσε αρκετά ε, γρήγορα. Ε, κατά τη γνώμη ή ε, στην αξιολόγησή του για την αξιοπιστία των λογαριασμών του 2008 το Συμβούλιο είπε ότι υπήρχαν προβλήματα και ενώ στα προηγούμενα έτη το Συμβούλιο θεώρησε ότι είχαν διαπιστωθεί σημαντικές αδυναμίες για το 2008 η γνώμη για την νομιμότητα των ε, συναλλαγών τονίζεται διότι το Συμβούλιο διαπίστωσε πολλές ε, ε, παράτυπες, παράτυπους διαγωνισμούς για συμβούλους παραβίαση των διοικητικών και δημοσιονομικών κανόνων και ε, όσον αφορά τώρα την Frontex. Η δήλωση του 2008 του ε, ελεκτικού συνεδρίου ε, θεωρεί ότι τα στοιχεία δεν είναι αξιόπιστα διότι υπήρξε μία μεταφορά 3,3 ε, εκατομμυρίων ε, ε, ποσών τα οποία μεταφέρθηκαν από την προηγούμενη χρονιά στην επόμενη ενώ 13 εκατομμύρια ευρώ καταργήθησαν συγχρόνως όμως ο προϋπολογισμός του οργανισμού αυξήθηκε κατά 29 εκατομμύρια ευρώ ή 69% σε σχέση με το παρελθόν έτος. Το επίπεδο αυτών των ποσών αποδεικνύει ότι η Frontex δεν είχε τη δυνατότητα να διεκπαιρεώσει το, τη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού της και ε, χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι οι οποίες δεν ε, καλύπτονται από τον κανονισμό του γραφείου και το θέμα συζητήθηκε με την Frontex. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι το ελεγκτικό συνέδριο διαπίστωσε ότι υπήρξαν βελτιώσεις εις ε, την απόδοση ε, των διαφόρων οργανισμών αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη ορισμένες ελλείψεις τις οποίες πρέπει να συζητήσουμε με τους οργανισμούς και τις εμπλεκόμενες, εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα όπως παραδείγματος χάρη να, να βρεθεί μια απλοποιημένη λογιστική να μπορέσουν να υπάρξουν περισσότερα εργαλεία ε, ε, αναφοράς που να βασίζονται στα αποτελέσματα και να προσφέρονται επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη συμβολή τους ή στην εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ενώσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Επιτροπή και τους οργανισμούς αυτούς για τη συνεργασία τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ε, να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να τελειώσουμε στις 6 και 4. Να δώσουμε λοιπόν ε, το λόγο στην εισηγήτρια. Σας παρακαλώ όλους να είστε πάρα πάρα πολύ σύντομοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Σαντάλοβα για ε, την εξαιρετική της εργασία θα αναφερθώ κατευθείαν στον κύριο Γκάρενσον ο οποίος είναι υπεύθυνο της ΣΕΠΟΛ και καταρχήν αναφέρομαι εις δαπάνε ε, ε, δαπάνες για την οργάνωση των σεμιναρίων που είναι ε, περίπου 60% των λειτουργικών δαπανών του οργάνου. Μου εξηγείτε γιατί δεν υπάρχουν δικαιολογητικά. Γιατί υπάρχουν υπάρχουν ε, αλλαγές ε, από την ε, αρχή του 2008 και από την εφαρμογή του συστήματος ABAC γιατί ε, ε, δεν ε, προσαρμοστήκατε στις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου από τον Ιούνιο του 2008 σχετικά με την κατακύρωση των, των διαγωνισμών. Τι έχετε να πείτε σχετικά με τον τρόπο διακηρύξεως δημοσίων διαγωνισμών διότι το, το ελεκτικό συνέδριο ε, διατυπώνει ανησυχίες. Δεν βλέπω να τις ε, ε, καλύπτεται. Σχετικά με την Όλαφ, το 2008 ξεκίνησε μία εσωτερική έρευνα για το έτος 2007 πώς αντιδράτε σχετικά με την έρευνα αυτή, συνεργάζεστε και σχετικά με τους πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για ιδιωτικούς στόχους για το 2007 μπορείτε να, ε, μπορείτε να μας πείτε τι έγινε με ε, τον έλεγχο από εξωτερική υπηρεσία θα ήθελα ο εκπρόσωπος της Όλαφ να μας πει τι γίνεται με την έρευνα η οποία διεξάγεται Όσον αφορά τις προσλήψεις, έχουν έχετε δυσκολίες προσλήψεων και φαντάζομαι ότι πρόκειται για, μια, διαρθρωτική, για ένα διαρθρωτικό πρόβλημα που οφείλεται στην θέση του κολεγίου στο Μπραμχιλ 70 χιλιόμετρα από το κέντρο Λονδίνου χωρίς να υπάρχει καλό μέσο μεταφοράς. Ε, σκοπεύετε να λύσετε το πρόβλημά σας. Ε, επίσης βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος ε, καταγραφής για τις κινητοποίησεις. Σχετικά με τον έλεγχο, ο Διευθυντής του Κολεγίου πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 5 να προσφέρει εις τον υπεύθυνο για την απαλλαγή μία έκθεση που να περιλαμβάνει ε, τις απαντήσεις στις συστάσεις του εσωτερικού ελεγκτή. Γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί ε, δεν ε, αναφέρατε τι, τις απαντήσεις σας σχετικά με τις συστάσεις που είχαν γίνει. Τώρα θα αναφερθώ στον υπεύθυνο της Frontex για τη διαχείριση του προϋπολογισμού. Σας ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη που, ζητώ συγγνώμη που διακόπτω. Ε, η τεχνική που θα ακολουθήσουμε είναι ερώτηση απάντηση. Τώρα κάνετε ήδη 12 ερωτήσει. Τι να κάνουμε. Να, να ακούσουμε την απάντηση. Διαφορετικά θα έχουμε ακούσει μόνο ερωτήσει και καμιά απάντηση. Ε, αυτό είχαμε πει σε την διαδικασία. Ερώτηση, απάντηση, ερώτηση, απάντηση. Για να ακούσουμε και κάποιε απαντήσει στι πρώτε ερωτήσει αυτέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ το Ελληνικό Συνέδριο για την υποστήριξή τους και για τον έλεγχο. Πάντως αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ του 2007 και του 2008 και ότι αλλάξαμε και το προσωπικό εντελώς. Οι ερωτήσεις τώρα για το κόστος των ε, μαθημάτων και των σεμιναρίων. Όταν έγινε η εισαγωγή του συστήματος και πέρασαμε το ένα σύστημα στο άλλο, είχαμε 6 άτομα προσωπικό. Ε, συγγνώμη, 8, 8, 8 άτομα προσωπικό για 100 διαφορετικές δραστηριότητες στα κράτη-μέλη. Ε, δεν ήταν εύκολο να τα κάνουμε όλα αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Αυτό ήταν το 2007 και σε ένα μεγάλο βαθμό και στο 2008. Πριν έχουμε την σημερινή κατάσταση όπου άλλαξε το προσωπικό, έχουμε νέο υπεύθυνο για τα λογιστικά, ένα νέο επικεφαλή της διοίκησης, νέος για τις προμήθειες που δεν τα είχαμε πριν. Πέρυσι, τον Ιανουάριο, όταν συναντηθήκαμε εδώ, είχε τελειώσει η χρονιά Το 2008 λοιπόν, γιατί αυτό συζητάμε, είχε λήξει ήδη. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για το έτος αυτό, αλλά μπορούσαμε και κάναμε πολλά για το 2009. Και αυτό είπα πέρυσι. Η απαλλαγή έρχεται ένα χρόνο μετά. Και δεν είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, διορθώσεις. Τώρα έρχομαι στις ερωτήσεις με τη σειρά μαθήματα και σεμινάρια. Τα οργανώνουν τα κράτη-μέλη με διάφορους εθνικούς κανόνες. Όταν εφάρμοσαν τους νέους κανόνες στα μέσα του 2008, δεν ήταν εύκολο ούτε εμείς, ούτε τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν απόλυτα. Το ηλεκτρικό συνέδριο έλεγξε για το πρώτο εξάμεινο του 2008 και το σύγκρινα με το δεύτερο εξάμεινο του 2008 και διαπίστωσε εξελίξεις. Και εμείς προσπαθήσαμε και τα κράτη προσπάθησαν. Τα κράτη δίνουν όλα τα οικονομικά έγγραφα, τα κείμενα, μετά την, το μάθημα του σεμινάριο. Εμείς λοιπόν πρέπει να συνεργαστούμε τα κράτη-μέλη δεν είναι εύκολο. Χρειάστηκε χρόνος γι' αυτό. Αν δείτε όμως τις ε, παράτυπες πληρωμές έχουμε μεγάλες διαφορές σε σχέση με το 2007. Για μαθήματα και σεμινάρια λοιπόν ίσως να υπάρξουν και στο μέλλον δυσκολίες. Παράδειγμα, τα κράτη-μέλη παίρνουν το δελτίο εισόδου ε, στα αεροπλάνα κλπ. Και δεν έχουν το δικαίωμα να μας στείλουν τα στοιχεία αυτά σε εμά. Εμείς δεν έχουμε λοιπόν τα στοιχεία αυτά. Μπορούμε να πάρουμε αντίγραφα, επίσημα αντίγραφα, μπορούμε να πάρουμε ένα σημείωμα, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα υλικά που εμείς δεν τα παίρνουμε στα χέρια μας στην περίπτωση που τα οργανώνει τα κράτη-μέλη. Αν επαναλαμβάνω συγκρίνουμε το 2007, το 2008 και το 2009, θα δείτε ότι το σύστημα ABAX με τους νέους κανόνες είχαμε σημαντική αλλαγή. Έτσι προμήθειες. Είχαμε περίπου 15 διαγωνισμούς ε, Καναδιό ήταν πολύ μεγάλοι όμω. Το πιο μεγάλο ήταν για την εκπαίδευση για το ABAC. Αυτό το κάναμε με την αρμόδια εταιρεία που παρέχει τις συμβουλές με συμβόλαιο με την Επιτροπή. Εμείς ζήσαμε περισσότερη εκπαίδευση, δεν αρκούσε αυτή που είχαμε ως τότε. Τελικά ζητήσαμε ένα επιπλέον συμβόλαιο στο τέλος του χρόνου. Και αυτό το συμβόλαιο το ηλεκτρικό συνάδειο λέει θα έπρεπε να είναι σε διαδικασία με διαγωνισμό και να μην χρησιμοποιηθεί το συμβόλαιο που ήδη έτρεχε. Δεν έχουμε ανοιχτό διαγωνισμό. Αυτό ήταν μια συνέχεια συμβολέου που ήδη υπήρχε με τη συγκεκριμένη αυτή εταιρεία συμβούλων. Πρέπει να το πω αυτό, γιατί ή άλλη προμήθεια διαγωνισμό που αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου δεν υπέστη καμία κριτική εκ μέρου του συνεδρίου. Προσλήψεις. Δυσκολίες υπάρχουν. Έκανα ένα φοβερό λάθο πριν από τρία-τέσσερα χρόνια που δέχτηκα ότι προσωπικό μπορεί να μεταφέρεται δωρεάν από κολέγιο στο αεροδρόμιο του Χίθρο. Η Όλαφ ε, ερεύνησε το θέμα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια υπέρ του προσωπικού. Τότε που το καταλάβαμε αυτό, με το που το καταλάβαμε το σταματήσαμε και ζητήσαμε να επιστραφούν τα χρήματα αυτά από τα πρόσωπα που είχαν χρησιμοποιήσει το σύστημα. Ανακτήσαμε τα χρήματα από όλους εκτός από έναν. Ε, τεχνικά δεν μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό, να πάρουμε τα λεφτά πίσω από το συγκεκριμένο πρόσωπο και λυπάμαι για το ότι κακώς πάρθηκε αυτή η απόφαση από εμά. Δεν το έκανα όμως επειδή ήθελα να χρησιμοποιήσω τα χρήματα της Ένωσης. Ήθελα να υποστηρίξω προσωπικό που δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει δημόσια μέσα μεταφοράς στη συγκεκριμένη διαδρομή. Μας κυνηγάει αυτό από πίσω δύο χρόνια τώρα. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, το σταματήσαμε. Τη μέρα που διαπιστώθηκε ότι ήταν λάθος και επαναλαμβάνω ε, μας επιστράφησαν όλα τα χρήματα με εξαίρεση ενώ από ένα πρόσωπο. Μετάνιωσα που πήρα αυτή την απόφαση, αλλά την πήρα. σταθερά στοιχεία ενεργητικού. Σωστά μας επέκρινε το συνέδριο ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού δεν είναι πάγια. <clears throat> Μέχρι το 2007 είχαμε ένα νέο σύστημα στοιχείων ενεργητικού <clears throat> και έχουμε δύο μητρώα αυτή τη στιγμή <clears throat> και για έλεγχο. Για έλεγχο και για λειτουργία. Το 2008 δεν χάσαμε τίποτα. Δύο πράγματα μόνο. Το έχουμε και στα δύο Μητρώα. Το ένα είναι τα, τα πάγια στοιχεία ενεργητικού. Εξακολουθούμε να έχουμε τα δύο συστήματα. Τίποτα δεν χάθηκε όμως. όσον αφορά τους ε, υπολογιστές, εκεί υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που είναι και στα δύο μητρώα και στα δύο συστήματα. Τώρα για το ίδιο το σύστημα. Στις 15 Ιανουαρίου πέρυσι εισήχθη το σύστημα Who Label. Όχι το 2008 που αυτή τη στιγμή είναι αντικείμενο ελέγχου λύθηκε αλλά δεν λύθηκε το Δεκέμβριο του 2008 λύθηκε τον Ιανουάριο του 2009. για την ε, έρευνα που έκανε η Όλαφ. Πληροφορήθηκα ότι έληξε, περατώθηκε αυτή η έρευνα και θα στείλουν έκθεση στον επικεφαλή του Διοικητικού Συμβουλίου. Την έκθεση αυτή δεν την έχω δει. Δεν ξέρω τι λέει. Αυτό είναι μια πάγια τακτική τη ε, όλα. Αυτό στέλνει την έκθεση και στην Κομισιόν στην Επιτροπή και στην Επικεφαλή του Δικαιωτικού Συμβουλίου. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ακόμα την έκθεση στα χέρια μου. Εγώ τουλάχιστον. Ούτε πληροφορίε. Ελπίζω να απάντησα σε όλε τι ερωτήσει. Πρόεδρος, επειδή ο χρόνος τρέχει, σας παρακαλώ να, απαντήτα, να απαντάτε σύντομα και κυρίως να δώσετε γραπτή απάντηση στα ερωτήματα. Δηλαδή, τις ερωτήσεις αδερφού Ματιέ προς την Όλαφ, παρακαλώ την Όλαφ να απαντήσει γραπτά. Γιατί 7 λεπτά έχουν μείνει και πρέπει να ασχοληθούμε με την Frontex και παρακαλώ να τεθούν οι ερωτήσεις για το Frontex. Πρέπει να πω όμω στον διευθυντή του ΣΕΠΟΛ ότι οι απαντήσει του δεν είναι καθόλου ικανοποιητικέ. Και ελπίζω να μα δώσει στη συνέχεια πιο συγκεκριμένε απαντήσει ε, γραπτά. Όσον αφορά τώρα τον διευθυντή τη Frontex, ιδιαίτερα όσον αφορά την διαχείριση του προπολογισμού. Ο προπολογισμό της ε, Frontex ε, αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια και ε, το Κοινοβούλιο και το 2006-2007 αλλά και για το 2008 ένα υψηλό επίπεδο μεταφορών και ακυρώσεων. Να μην σα αναφέρω ε, τα αριθμητικά στοιχεία, τα ανέφερε ήδη η κυρία Σαντόλοβα. Η ερώτησή μου είναι πώ ερμηνεύεται αυτή την κατάσταση που χαρακτηρίζεται από τόσο υψηλό επίπεδο ακυρώσεων και μεταφορών. Θα ήθελα συνέχεια να μου πείτε το πώ προβλέπετε ε, να αντιμετωπίσετε τι μελλοντικέ αυξήσει του προπολογισμού. Όσον αφορά τώρα τι επιδοτήσει. Ε, ε, δώσατε πάνω από γύρω στα 17 εκατομμύρια ευρώ με βάση μονομερείς αποφάσεις για επιδότηση που υπέγραψε μόνο ε, το Frontex. Όμως οι κανόνες που ισχύουν για τους οργανισμούς δεν προβλέπουν τέτοιου είδους μέσα. Πώς εξηγείται αυτή η κατάσταση ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επιδότηση ενός τέτοιου ποσού το σύστημα που παραθέτεται στις απαντήσεις σας και που θα έπρεπε να αρχίσει να ισχύει από τα μέσα του 2009 είναι λειτουργικό. Οι απαντήσεις του οργανισμού παραπέμπουν σε εξαιρετικές περιστάσεις που, ε, που οδήγησαν ε, στην επιδότηση. Αλλά ο αριθμό των εξαιρέσεων είναι υψηλό και το πρόβλημα αυτό ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη προπολογιστική διαδικασία. Ε, οπότε, ρωτώ, τα μέτρα τα οποία λήφθησαν από τον οργανισμό δεν είναι επαρκή. Όσον αφορά τώρα το Ταμείο, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνέταξε ο συνάδελφό μου Κριστόφ Φιενέλ για την ε, εκτέλεση του προπολογισμού του Frontex 2007 αναφέρει ε, απουσία πολιτική διαχείριση του Ταμείου. Τι γίνεται με το ζήτημα αυτό. Τέλο, όσον αφορά τη συνεργασία με τα κρατημέλη, θα ήθελα να αναφερθούμε σε ένα κρίσιμη σημασία στοιχείο που αφορά τη, λειτουργία του Frontex. Αναφέρομαι στη συνεργασία με τα κρατημέλη. Ε, Πώ επηρεάζει αυτή η συνεργασία την εκτέλεση του προπολογισμού και έχουν ληφθεί μέτρα για βελτίωση τη κατάσταση. Ευχαριστώ να θέλω την απάντησή σου στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Ευχαριστούμε. Πριν δώσουμε το λόγο στον από του Frontex, Καλό και τη ΣΕΠΟΛ και την Όλαφ και το Frontex, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε 4-5 λεπτά δεν μπορείτε να καλύψετε όλε τι ερωτήσει. Σα καλώ λοιπόν να μα δώσετε γραπτά τι απαντήσει σα σε βάθο μέχρι την 29η Ιανουαρίου, την Παρασκευή. Έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Chairman. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την Επιτροπή σας και στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο για την εξαιρετική σφίση συνεργασία. Μεταξύ μας δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ ε, σε ακρόαση ενώπιόν σας. Για λόγους ε, που είναι προφανείς και νομίζω ότι τα ζητήματα τα οποία ετέθησαν από την συγκήτρια είναι δικαιολογημένα. Ε, να ξεκινήσω ε, με την εξή υπενθύμηση. Η ευθύνη ε, του ελέγχου των συνόρων έγκυται στα κράτη-μέλη. Το Frontex συντονίζει τη συνεργασία στην περίπτωση που συμμετέχουν εθελοντικά τα κράτη-μέλη. Άρα, όταν εμείς αναπτύξαμε ε, την ικανότητα ε, του οργανισμού, ε, το κάναμε με βάση το εξή τρίγωνο. Η μία κορυφή του τριγώνου είναι η προθυμία των κρατών μελών, η άλλη κορυφή είναι η δημοσιονομική πόρη και η τρίτη η ανθρώπινη πόρη του Frontex και καταλαβαίνετε ότι τρεις αυτές κορυφές ε, συνυπάρχουν. Αν θέλουμε μόνο λοιπόν να αυξήσουμε ε, τους δημοσιονομικούς πόρους του Frontex και δεν από την άλλη δεν υπάρχει βούληση των κρατών μελών, τότε δεν πρόκειται ε, να να υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό το ένα. Δεύτερο, να σας πω ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός συνειδητοποίησης των προπολογιστικών ζητημάτων ε, που αφορούν τη χρηστή διαχείριση. Ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα. Ξέρουμε ε, το πρόβλημα στο οποίο αναφέρθηκε ε, και ε, ε, η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Έχουμε το πρόβλημα της έλλειψης τιμολογίων από τα κράτη-μέλη και βεβαίως το πρόβλημα της αναβολής ή ακύρωσης δραστηριοτήτων. Υπάρχουν βεβαίως λόγοι που εξηγούν την υπερβολική χρέωση, για παράδειγμα, όσον αφορά ε, θαλάσσιες επιχειρήσεις ή αεροπορικές επιχειρήσεις. εκεί δεν υπάρχει πρακτική δυνατότητα δραστηριότητα και, και πρέπει να δούμε το θέμα της επιστροφής. Τώρα, όσον αφορά τα τιμολόγια, από ό,τι υπολογίσαμε, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ από τότε που ξεκίνησε τις δραστηριότητε της στο Frontex αφορούν περιπτώσεις που δεν έστειλαν τιμολόγια ε, τα κράτη-μέλη. Πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για αυτό τα ποσό δεν έστειλαν τα τιμολόγια τους. Διότι ο κανόνας ήταν να είναι πολλά και ε, μικρής αξίας τα τιμολόγια. Και κατά την άποψή τους τα κράτη-μέλη δεν θεωρούσαν, και εδώ θα χρησιμοποιήσω τα λόγια των κρατών μελών, δεν, θεωρούσαν ότι άξιζε τον κόπο. Δηλαδή το όφελος δεν θα ήταν ανάλογο τη προσπάθεια για τόσο πολλά και μικρή αξία τιμολόγια. Βεβαίω. Όσον αφορά τον προπολογισμό του Frontex, όπως το 2007 και το 2008 αυξήθηκε κατά 3 εκατομμύρια ευρώ. Ε, μιλάμε δηλαδή για 35 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πάνω από το 1 τρίτο. Γιατί ο συνολικό προπολογισμό ήταν 70%. Και τι κάναμε λοιπόν με τα χρήματα αυτά. Αυξήσαμε την επιχειρη... τις επιχειρησιακές δραστηριότητες ε, του Frontex κατά 93%. Το ξαναλέω, 93% περισσότερο. αυξήθηκαν οι επιχειρήσεις όσον αφορά την εργασία μας. Οι μέρες κατάρτισης. Η αύξηση ήταν 192. Σχεδόν τριπλασιάσαμε τις ε, δραστηριότητες κατάρτισης με αυτά τα χρήματα. Πράγμα που σημαίνει ότι το πρόβλημά μας είναι διτό. Επειδή είχαμε αυτή την αύξηση κατά 30 εκατομμύρια ευρώ, όπως σας είπα, που έγινε στο δεύτερο εξάμεινο του έτους, δεν μπορούσαμε να προγραμματίσουμε και να ξεκινήσουμε τις δραστηριότητες που έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδότηση στο, σε εκείνο το οικονομικό έτος. Και ακριβώς για αυτό το λόγο η όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού, είχαμε ποσοστό 51%. Αλλά τώρα ε, τα νέα είναι καλά, γιατί μόλις πάρουμε τα κονδύλια που αφορούν τη μεταφορά από το 2008 στο 2009, το τελικό στάδιο υλοποίηση, εκτέλεσης του 2008 ε, ήταν ε, το, το τελικό ποσοστό ήταν 3%. Και εγώ αυτό το ποσοστό το θεωρώ καλό. Το πρόβλημα, όπως γνωρίζετε όμως, έχει να κάνει με το εξή. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει στο συγκεκριμένο φορολογικό έτος και όχι μέσω μεταφοράς. Η συγγήτρια ε, μας ε, αναφέρθηκε σε εξαιρέσει. Ναι, σωστό. Το 2008 είχαμε 167 εξαιρέσει. για πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Κυρίως λόγω της καθυστέρησης της τεκμηρίωσης από τα κράτη-μέλη. Αναφέρομαι στις θαλάσσιες επιχειρήσεις εμείς εσκεμμένα εστιάσαμε την προσοχή μας στα ζητήματα αυτά. Και ε, από ό,τι φαίνεται τα καλά νέα είναι το 2009 θα έχουμε μείωση του αριθμού των εξαιρέσεων ε, κατά το ίμιση. Και όσον αφορά την αξία αυτών των εξαιρέσεων θα μειωθεί κατά 85% και θα φτάσει μόλις στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τώρα, δύο λόγια πριν αναφερθώ στις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Για το 2009 να σας πω ότι ο βαθμός εκτέλεσης προπολογισμού ήταν 61%. Βελτίωση λοιπόν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Όπως σας είπα, είχαμε σημαντική βελτίωση ως προς τις εξαιρέσεις αυξήσαμε ε, την, την επιχειρησιακή ένταση και τις, κατά κατά 83% και τις ε, ε, ημέρες κατάρτισης που αυξήθηκε κατά 11%. Τώρα, ε, να σα πω το εξή. Ο τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να είναι περισσότερο δραστήρια όσον αφορά την επιχειρησιακή συνεργασία κυρίως μέσω ε, του, του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Για μας αυτό είναι ο βασικός τρόπος, το κλειδί για το πώς θα δεσμεύσουμε περισσότερο τα κράτη-μέλη για να είναι πιο ε, δραστήρια. Και πρέπει να σα πω ότι είχαμε θετικά αποτελέσματα και από άψη προπολογισμού. Τα 17 εκατομμύρια ευρώ ε, που Εδώ σε μονομερό. Εδώ να σα πω ότι οι εμπλεκόμενοι είναι ε, οργανισμοί ε, που προέρχονται από τι αρχές. Άρα εξορισμού είναι αξιόπιστη εταίροι. Ε, είχαμε μια κάπως διαφορετική ερμηνεία των δημοσιονομικών κανονισμών, τι μέσο δηλαδή είναι εφικτό και τι δεν είναι. Και αυτή τη στιγμή που όπως μας είπε και τόνισε ιδιαίτερα το ελεκτικό συνέδριο, να μην ακολουθήσουμε τη μονομερή οδό, θα, τα αλλάξαμε, αλλάξαμε τη διαδικασία και τώρα έχουμε ε, μια πολυμερή συμφωνία ε, που αφορά όλους πλην δύο. Εξαιρέσεις ήδη κάλυψε το ζήτημα αυτό όσον αφορά τη διαχειριστική πολιτική. Νομίζω ότι θα το... Ε, θα, θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες με τις γραπτές απαντήσεις, αλλά το ξαναείπα. Το 2008 ήταν πολύ καλύτερο από το 2007 και το 2009 ακόμα πιο καλό έναντι του το προηγούμενου έτους. Και αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι από ό,τι φαίνεται το ε, επίπεδο εκτέλεσης του προπολογισμού συνδέεται άμεσα, με το ποσοστό εκτέλεσης του προπολογισμού συνδέεται άμεσα με ε, το, το πόσο οριμάζει ο οργανισμός και η υπηρεσία μας. Σας ευχαριστούμε, περιμένουμε τις γραπτές παρατηρήσεις σας και επευθύνομαι και στην όλα. Και πριν πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσια διάταξη για ένα λεπτό να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο, ε, στην εκπρόσωπο του ελεκτικού συνεδρίου, την κυρία Σαντολόμπα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι το θέμα της χρήσεως μεγάλων αποφάσεων, δεν θε... αποφάσεων χορηγήσεων δεν είναι, ε, δεν είναι λανθασμένες ε, εφαρμογές. Είναι μέρος της νομικής ε, βάσης στην οποία βασίζονται οι Αποφάσισε. Ωραία, περνάμε τότε στο τελευταίο θέμα, στο σημείο 6 της ημερησίας διατάξεως. Με συγχωρείτε. Ε, με ενδιέφερε κάτι. Νομίζω ότι υπήρχε μία ερώτηση και για την Όλαφ. Δεν ξέρω εάν... Ε, ε, εάν ε, θα ήθελε και η Όλαφ να σχολιάσει διότι η Μεν Σέπολ ε, ε, σχολίασε. Το είπα ήδη, επειδή δεν έχουμε χρόνο, γιατί πρέπει να τελειώσουμε στι 6.30 και έχουμε και άλλο ένα ζήτημα στην ημερήσια διάταξη. Η Όλαφ θα απαντήσει γραπτά στην ερώτηση της εισηγήτριας μέχρι την 29η Ιανουαρίου. Τώρα, αν σε ένα λεπτό καταφέρετε να δώσετε μια απάντηση, να δώσουμε το, το λόγο στην Όλαφ. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα γραπτεί απάντηση. Ένα λεπτό έχετε το λόγο, έτσι για να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα μισή λεπτό αν είναι δυνατόν. Όντως νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω πολύ γρήγορα Όσον αφορά τη Frontex, καταρχήν δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Όσον αφορά την ΣΕΠΟΛ, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η έρευνα έγινε από την Όλαφ, ε, ξεκίνησε στις 19 Ιουνίου 2008 βάσει των στοιχείων οποία, τα οποία είχαν ε, σταλεί από την ΙΑΕΣ e και επιβεβαιώθηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο. Οι παρατυπίες που περιλαμβανόντουσαν και διαπιστώθηκαν και από την ΙΑΕΣ e και από το ελεγκτικό συνέδριο είναι γνωστές ότι τις βλέπω στο παράρτημα. Ο κύριος Ράντσον μας λέει ότι τα πράγματα βελτιωθήκανε αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι υπήρχαν πάρα πολλές παρατυπίες. Η εξέταση αυτή έγινε πάρα πολύ γρήγορα και πολύ δυναμικά για να καλυφθούν πολλές πιθανές παρατυπίες σε πολλούς τομείς ε, καταρχήν στο ενεργητικό, στα assets, στα procure procurement procedures ε, στις προσλήψεις, δηλαδή σχεδόν σε όλους τους κανόνες που αναφέρονται στη δημοσιονομική διαχείριση και ε, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή την 1η Δεκεμβρίου 2009 δηλαδή ολοκληρώσαμε αρκετά γρήγορα την έρευνα και ε, ο φάκελος αυτός έχει, έχει τώρα μεταβιβαστεί στους δικαιούχους δηλαδή καταρχήν τον τωρινό πρόεδρο της, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΟΛ, τον, ε, τους γενικούς γραμματείς ε, τον, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφού εμπλέκονται δημόσιοι υπάλληλοι και στις Βρετανικές αρχές. Δεν δίδεται στο κοινό ή σε άλλους και σας υπενθυμίζω ότι το, Όλαφ δεν είναι πειθαρχικό όργανο. Όταν ο κύριος Ράντσον θα προσεγγιστεί από τους ανωτέρους του θα μπορέσει είτε μπροστά στις δικαστικές αρχές ή στους ανωτέρους του να αμυνθεί βάσει των δικαιωμάτων του. Όντως η κατάσταση βελτιώνεται αλλά σας υπενθυμίζω ότι ο Όλαφ δεν είναι ελεγκτικό συνέδριο δεν είναι η δουλειά μας να πούν αν τα πράγματα κατουτερεύουν ή χειροτερεύουν απλώς να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν παρατυπίες εάν υπήρξαν και να τις υποδείξουμε όντως η βελτίωση υπάρχει αργά ε, υπάρχουν νέες διαδικασίες και ε, πέρυσι η απαλλαγή για την Όλαφ ε, νομίζουμε ότι σωστά πράξαμε διότι όλα εξελίσσονται θετικό. Σα είπα όμω ότι η έκθεση έχει ολοκληρωθεί και έχει σταλεί στους υπευθύνους. Περνάμε στο έκτο σημείο Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ζητήσει έκθεση 2008 και δίνω το λόγο στον κύριο Σλούμπορτ μέλο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Uh, uh, Ευχαριστώ. Διάβασα την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, σχέδιο έκθεσης μάλλον, του εισηγητή σας κύριο Ντόιτς. Συγχαίρω τον κύριο Ντόιτς. Καλύπτει όλα τα σημαντικά θέματα. ιδιαίτερα τα εξή τρία. Αναγνώριση της ανάγκης για εποπτεία των τραπεζών, η Ένωση να γίνει ο ένας από τους ε, μετόχους της τράπεζας, και το ότι το μέσον επένδυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης μπορεί να χρηματοδοτηθεί με χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Και εδώ πρέπει να δοθεί αυτή η απαλλαγή για αυτό το μέσο. Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, δεν θα πω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Πρώτα, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντόιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, όντως η ώρα είναι αρκετά προχωρημένη, γι' αυτό και θα ήθελα μέρου ε, μέρους ε, του Ουγγαρικού, Ουγγρικού Κοινοβουλίου να σας πω ένα ρητό όπου και εκεί τα πράγματα μέναν στην τελευταία στιγμή είχαμε ελάχιστο χρόνο να συζητήσουμε και τότε ο εισηγητής έλεγε πάντοτε ότι ε, τα κείμενα μιλούν ε, εύγλωτα και δεν χρειάζεται τίποτα να προσθέσουμε οπότε και εγώ το ίδιο θα πω δηλαδή ότι η αίτησή μου τα περιέχει όλα είναι όλα μέσα και οι κριτικές μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες της Επιτροπής ε, τον κύριο Μπράιαντ τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω γιατί πιστεύω ότι μας καλύψαν. Ο κύριος Χατζημαρκάκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως ο εισηγητής συνόψισε πολλά θέματα. Διαπιστώνω ότι υπάρχει πολύ έπαινος για την τράπεζα και όντως χαίρομαι διότι η τράπεζα έχει ακολουθήσει όλες τις συστάσεις μας μέχρι τούδε. Ένα θέμα μόνο το είναι το θέμα του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου και της αναπτυξιακής βοήθειας. Πρόκειται για χρήματα των φορολογουμένων που χρησιμοποιούνται ανεξέλεγκτα και θα ήθελα να προβλέψουμε να καλέσουμε εδώ μία κυβέρνηση, έναν υπουργό, το Συμβούλιο είναι αυτό και το γνωρίζουμε που προσπαθεί να ρυθμίσει ε, τα θέματα αυτά. Στη Γερμανία υπάρχει, ε, υπάρχει νέα κυβέρνηση όπου υπάρχει ένας ε, σωστός άνθρωπος τώρα ο οποίος ευχαρίστως θα έρθει εδώ να απολογηθεί και ευχαρίστως θα έπρεπε να τον προβλέψουμε το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα θα Ατεθεί το θέμα ε, διότι με τη συνθήκη της Λισαμπόνα τα θέματα αυτά αλλάζουν. Ευχαριστώ όμως τον εισηγητή. Όντως σχεδόν όλα τα θέματα υπάρχουν μέσα στην έκθεσή του. Ευχαριστώ κύριος Κάλφιν. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι όπως και στην έκθεση Deutsch υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή μας και έχουν σχέση με την εργασία αυτής της Επιτροπής. Δεν θέλω ε, να θίξω τα διάφορα θέματα που έχει αναφέρει και που είναι ενδιαφέροντα αλλά ο κύριος Καμπτωσίου είχε μια υπηρεσία που κλείνει τώρα και στις 15 ε, Φεβρουαρίου θα υπάρξει μια έκθεση σχετικά με το, τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επένδυσης η οποία θα συζητηθεί το Μάρτιο στην Επιτροπή μας διότι περιέχει πολλές ιδέες. Υπάρχουν λοιπόν πολλά θέματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα όπως και στην έκθεση του κυρίου Ντόιτς. Πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη μας την εργασία της ειδική Επιτροπής και όταν μιλάμε για το χρονοδιάγραμμα που θα υιοθετηθεί η έκθεση αυτή θα πρέπει να συντονιστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθούν όλα τα βασικά θέματα λόγω των διαφόρων λύσεων που μας έχουν προταθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ήβαν. Σα ευχαριστώ. σε αφορά το σχέδιο έκθεση του κύριου Ντόιτς, νομίζω θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθεί ε, στην ε, έκθεση που αφορά τα, πρόγραμμα, τα προγράμματα τεχνικής αρρωγής. Ε, γιατί πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να ενταχθούν να και τα νέα προγράμματα, τα νέα πενταετή προγράμματα και στα πλαίσια αυτά της οικονομικής κρίσης και της Ατζέντα Λισαβόνας η οποία μπήκε σε παρένθεση, αν θέλετε, ε, λόγω των, της οικονομικής κρίσης, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό αυτή η, ε, ε, η διευκόλυνση, η χρηματική διευκόλυνση και, το, και η κοινή ανάληψη του κινδύνου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της έρευνας και της καινοτομία. Ευχαριστώ, κύριος Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όσο... Ε, αυξάνεται η οικονομική κρίση στο μέλλον, θα πρέπει να βρούμε άλλου μηχανισμού για να χρηματοδοτήσουμε σημαντικά προγράμματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε καλά παραδείγματα, τον Τζέρεμι, τον Τζάσμιν και τον Τζέσικα. Και αν διαβάσετε την έκθεση, σελίδα 8, θα δείτε ότι τον Τζάσμιν και τον Τζέσικα και τον Τζέρεμι αναφέρονται στη συγκεκριμένη έκθεση. Και πραγματικά πρέπει να αναφερθείτε και στο, στη δυνατότητα να γίνει αξιολόγηση των μέσων αυτών στο μέλλον. Είναι εξαιρετικό αυτό το οποίο αναφέρεται. Αυτό όμω το οποίο δεν αναφέρεται είναι ότι ε, δεν αναφέρεστε ε, στο Τζέσικα, ε, γιατί είναι πολύ σημαντικό ο χρηματοδοτικό μηχανισμό που θα ξεκινήσει στο μέλλον. για παράδειγμα, η Ουαλία θα ξεκινήσει προ το τέλο του χρόνου μια πρωτοβουλία στα πλαίσια, στα πλαίσια του Τζέσικα. Άρα θα πρέπει να αξιολογηθούν και αυτέ οι προσπάθειε. Δεν μπορείτε να συμπεριλάβετε λοιπόν το Τζέσικα στην έκθεσή σα. Εκτό δηλαδή του Τζέρεμ και του Τζάσμιν, να συμπεριλάβετε και το Τζέσικα. Θέλετε να μιλήσετε κύριε Ντόιτ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και για τις συμβουλές τους και τις ε, απόψεις που διετύπωσαν ο πρόεδρος ήταν συνεπής και έτσι τελειώνουμε, ξεπεράσαμε το χρόνο μόνο τέσσερα λεπτά. Δεν θέλω να καταχρεστώ το χρόνο ούτε καν των διερμηνέων, διότι όλα τα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν πιστεύω ότι μπορούν να απαντηθούν. Δηλαδή, στις τροπολογίες θα λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα θέματα και θα τα περιλάβουμε. Είναι πολύ βασικό αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος δηλαδή πέραν της τωρινής εκθέσεως θα έπρεπε να λάβει κανείς υπόψη του και τις υπόλοιπες δραστηριότητες και να τις συντονίσει. Θα εξετάσουμε τι γίνεται ε, κατά την κατάρτιση της ε, τελικής μορφής της εκθέσεως αυτής και πιστεύω ότι χρησιμοποιώντας ε, τα συγκεκριμένα προγράμματα όταν η αποτελεσματικότητα ελέγχεται ή όταν ελέγχεται πώς πρέπει να συνεχιστούν συγκεκριμένα προγράμματα προγράμματα. Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη και θα καταρτιστούν τροπολογίες οι οποίες κατά τη συζήτηση ή στην Ολομέλεια θα μπορέσουν επίσης ε, να ε, περιληφθούν κατά τρόπον ώστε να ε, κλείσουμε αυτή τη διαδικασία στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 11 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο στις 3.30. Ευχαριστώ όλους.